Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση για την ασφάλεια των πληροφοριών και του διαδικτύου. Ευχαριστώ τον Άντριο Σβάπ, τον εισηγητή, πάρα πολύ που διοργάνωσε την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα και τα άλλα μέλη που παρίστανται και ιδιαίτερα καλωσορίζω τους ομιλητές που θα παρουσιάσει τα θέματα. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό. Ουσιαστικά σκοπός είναι να έχουμε ένα ευρύ φάσμα οπτικών γωνιών όσον αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και ήταν εισηγητής μας ο κύριος Σβάμπ. Χωρίς να καθυστερήσω, θα του δώσω τη δυνατότητα να κάνει μια εισαγωγή στην πρόταση. Πριν το κάνω αυτό, Καλωσορίζω οποιονδήποτε μας παρακολουθεί το διαδίκτυο. Έχουμε καμιά φορά πολύ μεγάλο ακροατήριο στο διαδίκτυο. Και καλώς ήρθατε λοιπόν, Καλωσορίζω ορίστε θεατές που παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Άντιους Σφαμπ, θα σου δώσω το λόγο να κάνεις μια παρουσίαση της πρότασης. Θα ήθελα να πω πώς θα εκτυλιχθεί η εκδήλωσή μας στο πρώτο κομμάτι της συνεδριάσεως μέχρι τις 4. Πρώτο θέμα, είναι πώς εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ασφαλείας των δικτύων και των πληροφοριών και μετά, στο δεύτερο τμήμα, από τις 4 μέχρι 5 παρα 5, κοινή αντίληψη της ασφαλείας στον κυβερνό χώρο, κάλυψη των κενών και χαίρομαι που έχουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες μαζί μας. Εν συντομία θα σας παρουσιάσω πριν πάρουν το λόγο, αλλά να σας πω ότι οι συμμετέχοντες, τα μέλη και στο κρατήριο το λέω αυτό, Υπάρχει βιογραφικό όλων των ανθρώπων που θα πάρουν το λόγο. Δεν θα διαβάσω δημόσια το βιογραφικό τους, μπορεί να διαβάσει κανείς, άμα ενδιαφέρεται, ξεχωριστά. Αυτά έχω να σας πω για την τυπική διαδικασία. Ο καθένας από τους ομιλητές μας έχει χρόνο συγκεκριμένο. Θα έχουν ένα ρολόι μπροστά τους για να τους βοηθά για το χρόνο. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τα χρονικά όρια, μπορούν τα μέλη μετά να θέσουν ερωτήσεις και ίσως να πάρουν το λόγο κι άλλοι και μετά θα στραφώ και προς το πάνελ το οποίο θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε διαδραστικό διάλογο ε, ερωταπαντήσεων. Λοιπόν, Άντιο Σβάμπ, θα σου δώσω το λόγο για μια σύντομη εισαγωγή της πρότασης και τι σχέδια έχεις για το θέμα και μετά θα προχωρήσουμε στην ακρόαση αυτή καθεαυτή. αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνει τη δυνατότητα να πω μερικά λόγια πριν ξεκινήσουμε την ακρόαση. Θα ήθελα εισαγωγικά, ουσιαστικά, καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία για το ότι οι συνεργάτες και συνεργάτες ε, με τέτοιες προσπάθειες συνεισέφεραν στην προπαρασκευή προετοιμασία αυτής της ακρόασης. Εμείς ως αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για αυτή την οδηγία για το δίκτυο και την ασφάλεια δικτύου στον κυβερνοχώρο σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή μια ολόκληρη σειρά άλλων θεμάτων μπορούμε να αποσαφηνίσουμε απόψε. Καταρχήν ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή είμαστε όπως καμιά άλλη επιτροπή σε θέση να πάμε σε εύρος, σε μεγάλο φάσμα το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε. Ολιστική προσέγγιση λέμε στον τίτλο ήδη. Στόχος πρέπει να είναι σε μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια να θέσουμε το ερώτημα σε ποιο βαθμό και σε ποιους τομείς ε, σήμερα στη ζωή μας η κυβερνοασφάλεια για τις καταναλώτριες και καταναλωτές είναι ένα θέμα που τους αφορά άμεσα. Ξεκινάμε το ερώτημα αν πρόκειται εδώ για εθελοντική δράση ή για δεσμευτική ρυθμιστική δράση για νομοθετικά μέτρα δηλαδή εθελούσιου εθελοντικού χαρακτήρα υποχρεωτικού. Μετά, ποια στοιχεία θεωρούμε ως κέρια στοιχεία υποδομής με τα οποία οι καταναλωτές καθημερινά έρχονται σε επαφή και που όλα σε ένα βαθμό αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και που δεν είναι τόσο ανθεκτικά όπως θα το ήθελαν οι περισσότεροι καταναλωτές ή πιστεύουν ότι είναι. Και το δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο τμήμα της ακρόασής μας ε, σήμερα το απόγευμα, φυσικά θα εξετάσουμε το θέμα με ποιο τρόπο εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να συνεισφέρουμε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την βελτιώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά τα διασυνοριακά θέματα και ζητήματα που αφενός ε, για την οδηγία αυτή για μας διαδραματίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο, αλλά και από την άλλη πλευρά οι βελτιώσει των ελάχιστων απαιτήσεων από τα κράτη-μέλη, πώ μπορούμε αυτά να τα θέσουμε στο επίκεντρο. Και ελπίζω ότι οι προσκεκλημένοι μας ε, αγορητέ σήμερα το απόγευμα θα μας προσφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες για να μας διαφωτίσουν. Το δεύτερο τμήμα του απογεύματος βρίσκεται υπό τον τίτλο «Τι μπορεί να κάνει μια κοινή κατανόηση» και τι μπορεί να είναι αυτή η κατανόηση για το ε, την προσέγγιση και κατανόηση του θέματος της κυβερνοασφάλειας. Προσβλέπω να ακούσω τις παρατηρήσεις στο δεύτερο πάνελ από τους αγορητές σήμερα το απόγευμα, πώς δηλαδή η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά μπορεί, μπορούν να βελτιωθούν. Που ναι με σήμερα με μια ολόκληρη σειρά κυβερνοεπιθέσεων βρίσκονται αντιμέτωποι, αλλά και που για τα θέματα των καταναλωτών γενικά, για την λειτουργία αυτής της αγοράς, ε, παρισφρέουν, αναμειγνύονται και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και χαίρομαι για το ότι οι επαΐοντες, ε, οι πραγματογνώμονες μπορούν να μας δώσουν αξιόλογα στοιχεία τα οποία εγώ ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εντάξω στην έκθεσή μου. Αδειμονώ να ακούσω τι έχουν να μα πούν οι πραγματογνώμονε σήμερα το απόγευμα. Υπαρκεί μέχρι εδώ λοιπόν αυτή η εισαγωγή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά α προχωρήσουμε στο πρώτο τμήμα τη ακροάσεω. Θέλουμε να ακούσουμε τι δικέ σα απόψει τι απόψει των εμπειρογνωμόνων. Πώ να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα δηλαδή, πώ θα εξασφαλίσουμε εξασφαλίσουμε, ίσω δεν είναι σωστή λέξη, δεν είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι και να εξασφαλίσουμε 100%, να έχουμε το ύψιστο δυνατό επίπεδο ασφαλεία όσον αφορά πληροφορίε στο διαδίκτυο και πώ βλέπετε την σημαντική αυτή πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε τρει διαφορετικέ απόψει. Πρώτα απ' όλα, Αριάν Κιζάου από το Κέντρο Ευρωπαϊκή Πολιτική, ανάλυτη πολιτική στον τομέα χρηματοστικών ε, υπηρεσιών, Έλενα Ράου, που είναι συντονίστρια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και Υπουργό ε, Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνία στην Εστονία, και εφόσον είναι στην κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη εμπειρία κυβερνοεπιθέσεων ε, όσον αφορά ένταση των σχέσεων και των προβλημάτων σε σχέση με το μέγεθος της χώρας και μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η εμπειρία σας και ξέρω ότι εργάζεστε για μια στρατηγική της χώρας σας για την Εστονία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πώς θα συμβάλλει η ευρωπαϊκή πρόταση στη γενική ασφάλεια και της χώρας. Και μεγάλη χαρά για πρώτη φορά, είχα τη χαρά να καλωσορίσω στην Επιτροπή μου κάποιον από πολύ ψηλό επίπεδο της Ευρωπόλ, τον Όλιβερ Μπέργκεστάικ, επικεφαλής της στρατηγικής και πρόληψης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος. Καθημερινά αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και αυτό νομίζω είναι κάτι που συμβάλλει στον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας δώσουμε, θα σας δώσουμε το πολύ ένα τέταρτο για να μιλήσετε, αλλά ε, εδώ η γραμματεία συνοφριώθηκε με αυτά που είπατε 10 λεπτά. Μπορώ να είμαι αρκετά ευέλικτο, αλλά θα θέλαμε να έχουμε και ρωτήσει που υποβληθούν. Ελπίζω να μην πρέπει να σας διακόψω. Αν δείχνετε διαφάνειες θα φαίνονται εκεί στις οθόνες και θα πάρετε και αντίγραφα των διαφανειών και στο διαδίκτυο νομίζω. Δεν ξέρω αν έχουμε πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας. Αν οι θεατές από το διαδίκτυο αν θα βλέπουν τις διαφάνειες. Φαίνεται ότι ναι. Εγώ δεν έχω την δυνατότητα να βλέπω τι κάνει δική μου επιτροπή, στη δική μου επιτροπή, αλλά ελπίζω ότι και οι θεατές βλέπουν τις διαφάνειες. Αριέν, σου δίνω το λόγο και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση Είμαι επιστημονικά υπεύθυνη για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Είναι μια δεξαμενή σκέψη ε, το, το δικό μας ε, Ίδρυμα. Αναλύουμε σημαντικά πολιτικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύσσουμε και στρατηγικές για την ευρωπαϊκή πολιτική πέρα από αυτά. Αυτά έχουν και την έκφρασή τους στο γεγονός ότι μια συνθήκη σύμβαση πλαισίου για την Επιτροπή ΕΚΟΝ εκπονούμε ε, εξυπηρετεί ε, κοινό όφελος και είμαστε ανεξάρτητοι από κόμματα ή από άλλους φορείς κύριο έργο μα είναι η αξιολόγηση οικονομική και νομική των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αξιολογηθούν οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε συνεντεύξεις ε, με του φορεί και αρμόδιου από του διάφορου τομεί. Με τη σημερινή πρόταση σε βάθος ε, ήρθαμε σε επαφή και εξετάσαμε τι πτυχέ αυτέ και θέλουμε να σα παρουσιάσουμε την αξιολόγηση αυτή. Στην δική μου παρουσίαση θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στην οικονομική αναγκαιότητα για μια κανονιστική παρέμβαση σύμβαση ε, για τις ε, αγορές ε, και τις δημόσιες αρχές. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο άρθρο 14 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αναφερθώ υπό ποιου όρους και προϋποθέσεις αυτά που προτείνονται ως διορίες για την αναφορά και καταχώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης και εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Πρώτον, για τις ε, απαιτήσεις για την ασφάλεια όσον αφορά τους συμμετέχοντες στις αγορές. Πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 14 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλοι αυτοί να υλοποιούν προδιαγραφές και ρήτρε για τα δίκτυα που θα ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη μορφή και ε, έκφραση της τεχνολογίας. Δηλαδή η χρήση όλων αυτών πρέπει νομικά να ρυθμίζεται. Έτσι ουσιαστικά παρεμβαίνουμε σημαντικά στην ελευθερία των ε, επιχειρήσεων. Όμως ε, ο στόχος είναι τα δίκτυα να καταστούν ανθεκτικότερα σε σχέση με επιθέσεις ή παρεμβάσεις εκ των έξω και να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας έτσι. Γιατί αυτό όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ένα ίδιο συμφέρον να προστατεύουν τα συμφέροντά τους σε αυτό το επίπεδο και να επενδύουν αρκετά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο. Όμως ε, για τους πολίτες κάτι τέτοιο δεν είναι άμεσα ε, ευδιάκριτο. Αν γίνει μια κυβερνοεπίθεση και γίνει μια διάρρηξη ή επέμβαση σε μια επιχείρηση στον κυβερνοχώρο, αυτό δεν, δεν γίνεται γνωστό σε όλους και το γεγονός γίνεται γνωστό μόνο όταν μέρη ή τμήματα του συστήματος δεν λειτουργούν απροβλημάτιστα ω συνήθως και παραμένει αδιάκρι, δυσδιάκριτο αυτό. Μόνο οι, πολ... οι πελάτες ε, υφίστανται τη ζημιά στο τέλος και στο τέλος τέλος με τα στοιχεία τους είναι εκείνοι που πληρώνουν τα σπασμένα. Είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να ταυτοποιηθεί μια επιχείρηση σε σχέση με τέτοιες επιθέσεις ε, κλοπών στοιχείων ή σε τέτοιου είδους ε, επεμβάσεις που έχουν υπάρξει. Δηλαδή οι συμμετέχοντες ε, στην αγορά δεν θα πρέπει λόγω της ελλειπούς ασφάλειας να συνεχίσουν να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο το γεγονός της ευθύνης ή υπευθυνότητας δεν λειτουργεί εδώ επαρκώς. Ναι, μεν μπορεί κανείς για παράδειγμα να διαπιστώσει την μη λειτουργία μιας υπηρεσίας και να αναφερθεί σε κάποια επιχείρηση, η απέτηση όμως αποζημίωσης συνεπάγεται τέτοιες δυσκολίες λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων που πολύ δύσκολα μπορεί να διακριβωθεί. Συνέπεια είναι ότι δεν έχουν επαρκή ευθύνη οι επιχειρήσεις και δεν γίνονται οι αναγκαίες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Μια και η αρχή λοιπόν της ευθύνης ή της υπευθυνότητας δεν αρκεί, μια ρυθμιστική επέμβαση είναι αναγκαία. Γι' αυτό οι τεχνικές απαιτήσεις στο άρθρο 14 είναι νόμιμες και σκόπιμες. Τώρα αυτά που προτείνονται ως διορίες για την καταχώρηση ως προθεσμίες στο 14 θέλω να τα εξετάσουμε και να δούμε αν αυτά υπαρκούν ώστε η ανθεκτικότητα των δικτύων και των ε, συστημάτων πληροφορικής να μπορούν να καλυφθούν. Οι συνεντεύξει με του εμπλεκόμενου μα έδωσαν ε, ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Βρήκαμε ότι ήδη τώρα πολλέ επιχειρήσει, όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια σε εθελούσια βάση άτυπα συνεργάζονται μεταξύ του. Οι επιχειρήσει συνεργάζονται μεταξύ του με ανταλλαγή πληροφοριών για τι πιο σημαντικέ τέτοιε περιπτώσει ασφάλεια. Όμω, το πιο σημαντικό είναι ότι ανταλλάσσουν απόψει για λύσει και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Αυτέ οι ανταλλαγέ πληροφοριών οδηγούν ώστε τα δίκτυα από αμφότερους τους εταίρους να μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικά και πιο ασφαλή. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Μια ενεργειακή επιχείρηση συνεργάζεται με έναν ομόλογο στο εξωτερικό, με ένα ομόλογο ίδρυμα. Θέλουν να βρουν οι επιχειρήσει ποιε περιπτώσει ασφάλεια απασχολούν αυτή τη στιγμή τα δίκτυα αυτά. Υπάρχει ελπίδα από, από τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις να γνωρίσουν έγκαιρα τα σχετικά προτού συμβεί ζημιά στις ίδιες αυτές επιχειρήσεις. Μέσω λοιπόν της συνεργασίας αυτής και του συντονισμού ελπίζουν να κερδίσουν χρόνο ώστε να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπρος Είδαμε λοιπόν ότι τέτοιου είδου συνεργασίες στο μεγαλύτερο βαθμό μέσα σε έναν ίδιο τομέα ή κλάδο διεξάγονται. Μια και ένας ίδιος τομέας ή κλάδο χρησιμοποιεί το ίδιο λογισμικό τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό οι επιχειρήσει αυτές σε ίδιο επίπεδο μπορούν να κινηθούν και με το ίδιο αυτό επίπεδο μπορούν να ε, προβληματιστούν στην ανταλλαγή απόψεών τους για να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα προβλήματα. Σκεφτήκαμε μετά πώς μπορούν τα κυριότερα θέματα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια να τυποποιηθούν ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πρόγνωση. Μια πρόγνωση πρόβλεψη αν η εθελούσια αυτή δράση επαρκεί ώστε να διασφαλιστεί πανευρωπαϊκά μια ασφάλεια σε αυτά τα δίκτυα. Υπό ποιου όρου και προποθέσει και πότε εθελοντικά θα, συνεργάζονται οι επιχειρήσει αυτέ και θα ανταλλάσσουν πληροφορίε για τέτοιου είδου περιστατικά περιπτώσει ασφάλεια η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι σχετικά σαφή. Συνεργάζονται οι επιχειρήσει όταν από αυτή την συνεργασία προσδοκούν μια πρόσθετη αξία. Δηλαδή ένα είδο πριμ ή μπόνους που μέσω αυτής της πρόσθετης συνεργασίας διασφαλίζεται. Αυτή η πρόσθετη αξία είναι, α το πω έτσι, η θετική επίπτωση από αυτή τη συνεργασία για αμφότερους του εταίρους στο πλαίσιο αυτή τη συνεργασία. Αν την πρόσθετη αξία νομισματικά, οικονομικά θέλει κανείς να αξιολογήσει, αυτή η πρόσθετη αξία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το εξοικονομηθέν κόστος ε, για την αντιμετώπιση των ζημιών ε, στο δίκτυο από κυβερνοεπιθέσεις ή το εξοικονομηθέν κόστος ε, από δράσεις στην αγορά έναντι των πελατών για να ανακτηθεί το απολεσθέν κύρος. Αυτό ήδη μπορεί να είναι αρκετό και να καλύπτει την δυνατότητα να υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Συνεργασία και πρόληψη είναι σημαντικά στοιχεία αυτής της προληπτικής δράσης της δαπάνης εκατομμυρίων κονδυλίων για να ανακτηθεί η απολεστήσα εμπιστοσύνη σε σχέση με πελάτες. Αναφέρομαι στο γεγονός σε σχέση με την εταιρεία Sony το 2011. Τεράστια κονδύλια απαιτήθηκαν από τη Sony ώστε να ανακτηθεί η απολεστήσα εμπιστοσύνη λόγω του τροθέντος κύρους της Sony από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Μια και τα τροτά σημεία μέσω αυτής της συνεργασίας μπορούν ταχύτερα να εντοπιστούν και να αρθούν να αντιμετωπιστούν με τέτοιου είδου συνεργασίες όταν και τα δύο τμήματα και οι δύο εταίροι υπόσχονται για τον εαυτό τους ένα τέτοιο κέρδος ως πρόσθετη αξία είναι θετικά γεγονότα. Και όταν γίνεται μια τέτοια, όταν λειτουργεί μια τέτοια συνεργασία καταλήγουμε σε ένα υψηλότερο βαθμό ασφάλεια έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό έχει ε, υπαρξιακό χαρακτήρα, αλλά η περαιτέρω διάθεση μόνο πάλι μέσω συνεργασία μπορεί να διασφαλιστεί. Για το αρχικό ερώτημα, επαρκεί η εθελούσια αυτή η ρύθμιση, ώστε στα δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο ασφάλεια. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, έχουμε τη συνεργασία των διαθροτικών ταμείων σε, που αναλύσαμε σε εθελοντική βάση και αυτό και να δώσουμε απάντηση πότε, ποιε επιχειρήσει και γιατί συνεργάζονται μεταξύ του. Διαπιστώσαμε ότι η εθελούσια τέτοια συνεργασία ε, υλοποιείται όταν τρία κριτήρια υλοποιούνται. Πρώτον, πρέπει αξιολογήσιμα τέτοια στοιχεία και συγκρίσιμα να μπορούν να απορρέουν ως στοιχεία. Χρειάζονται επιχειρήσεις στοιχεία με τη βοήθεια των οποίων τα δίκτυά τους μπορούν να προστατευτούν εναντί τέτοιων ε, επιθέσεων. Δηλαδή πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου αυτές οι πληροφορίες ώστε να συνεισφέρουν αυτόματα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένες λοιπόν και στοχοθετημένες αυτές οι πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ξεκινήσει βήματα και διαβήματα μια τέτοια επιχείρηση για την αντιμετώπιση κολλημάτων και προβλημάτων. Ροή πληροφοριών το δυνατόν ταχύτερο, ταχύτερα πρέπει να διασφαλίζεται για να αποφευθούν ζημιές ή το ταχύτερο να μπορέσουν να αποκατασταθούν. Και τρίτον, εμπιστοσύνη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βέβαιες και να διασφαλίζεται ότι με ε, εχεμήθεια θα διασφαλίζεται ο απόρριτος χαρακτήρας αυτών των στοιχείων, ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας για να αποφύγουν ζημιές. Αυτά τα κριτήρια είναι σημαντικά. Δηλαδή αξιολογήσιμες ε, εξειδικευμένες πληροφορίες, ροή πληροφοριών και σε εθελοντική βάση συνεργασία και εχεμήθεια, ε, αν δεν υλοποιείται ένας ε, από αυτούς τους παράγοντες επαρκώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί συνολικά μια αποτελεσματική συνεργασία. Απορρέει το συμπέρασμα ότι μια εθελοντική συνεργασία μόνο μεταξύ κάποιων λίγων εταίρων ή ομολόγων θα γίνεται που ένας έχει εμπιστοσύνη στον άλλον και δίνουν στοχοθετημένα εξειδικευμένες πληροφορίες ο ένας τον άλλον. Από αυτήν την παρατήρηση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εκείνοι οι οποίοι καταλήγουν σε μικρότερα πλαίσια συνεργασίας, δηλαδή διακλαδικά ε, ή τομεακά, εκεί ε, εντοπίζονται τα προβλήματα. Υπό τον εθελοντικό χαρακτήρα δεν είναι δημόσια αυτά τα στοιχεία, παραμένουν μεταξύ των εταίρων της συνεργασίας. Για να μπορέσει όμως σε μεγάλο βαθμό, σε όλο το επίπεδο, σε όλο το φάσμα δράσης να βελτιωθεί η ασφάλεια στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, πρέπει το δυνατόν περισσότεροι να μπορούν να συμμετέχουν. Όσο μεγαλύτερο το εύρος, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα της συνεργασίας. Συνοψίζω η ανάλυση τη της συμπεριφοράς συνεργασίας όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας των δικτύων για την κυβερνοασφάλεια δείχνει ότι η ε, εθελοντική συνεργασία μόνο σε μικρό βαθμό και ε, ενδοτομεακά ή ενδοκλαδικά ε, μπορεί να διεξάγεται με αυτή τη μορφή. Η πανευρωπαϊκή προσέγγιση δεν διασφαλίζεται. Για να διασφαλίσουμε, διασφαλίσουμε όμως ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας θα πρέπει πολύ μεγαλύτερο εύρος συνεργασίας να διασφαλίζεται. Μια και έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από την ηλεκτρονική ροή πληροφοριών στην οικονομία και έχουμε και όλο και περισσότερους κινδύνους στους οποίους εκτιθέμεθα στον κυβερνοχώρο. Για την ελεύθερη συνεργασία, ε, εθελοντική συνεργασία σημαίνει ότι ένας ε, χαρακτήρας ε, καταχώρησης θα πρέπει να διασφαλιστεί ώστε σε εθελοντική βάση όσοι συνεργάζονται να καλύπτονται όσον αφορά την ασφάλειά τους στο μεγαλύτερο εύρος. Οι πληροφορίες θα πρέπει από όλους να είναι διαθέσιμες για όλους. Τότε όλοι οι συμμετέχοντες εξ ιδίου συμφέροντος θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίε ώστε να καταλήξουν σε IT ασφάλεια. Και εδώ ακριβώς έχουμε το πρόβλημα της εθελοντικής τώρα χρήσης και λειτουργίας. Μια και όλα τα συλλεγέντα στοιχεία από αυτές τις καταχωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμεσα και άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους, έχουν ένα χαρακτήρα δημόσιου αγαθού. Σαν συνέπεια έχουμε ένα πρόβλημα λαθρεπιβατών, free riding. Όλοι θέλουν αυτές τις πληροφορίες και θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν, κανένας όμως δεν θέλει να τις δίνει ο ίδιος. Και δυνάμει να εκτίθεται και φυσικά δεν θέλει και να πληρώνει τέλη, ε, εισφορές ε, και, ε, και δαπάνες να καλύπτει. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος λαθρεπιβατών, οι προτάσεις για την καταχώρηση όσον αφορά τέτοια συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια είναι σκόπιμα και εξυπηρετούν τους στόχους. Εκείνο το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας διασφαλίζεται που με θελοντικό τρόπο δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Οι προθεσμίες και διορίες οδηγούν ώστε επιχειρήσεις τέτοιου είδους πληροφορίες για σημαντικά θέματα ασφάλειας να μπορούν να τα γνωστοποιούν. Έτσι, στην υπηρεσία, αρμόδια υπηρεσία μπορεί να υπάρξει μια βάση δεδομένων και μια εικόνα συμβάντων. Από αυτή την εικόνα συμβάντων και βάση δεδομένων μπορεί να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί ο κίνδυνος και το συμβάν. Έτσι πρέπει να διασφαλίσουμε όμως ότι οι διορίες και προθεσμίες δεν θα χρησιμοποιείται ώστε να συλλέγουμε περιτά στοιχεία και να έχουμε μια συσσόρευση περιττών στοιχείων πολύ περισσότερο στη διατύπωση του άρθρου 14 πρέπει με αυτή τη διαδικασία σκοπ εξειδικευμένα χρήσιμα στοιχεία να συλλέγονται για τις προθεσμίες και διαδικασίες είναι σημαντικό οι αρχές αυτές που αναφέραμε για τη συνεργασία να είναι σεβαστές. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα και μόνο τότε υπάρχει αρκετή αποδοχή από τους οικονομικούς κύκλους. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 14. Οι διαδικασίες είναι αναγκαίες ώστε να έχουμε μια βάση δεδομένων για την αντιμετώπιση κυβερνοσυμβάντων ε, στο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας. Πολύ πιο σημαντική είναι όμως η συνεργασία με αυτούς τους φορείς και υπηρεσίες. Πρέπει να μπορούμε να δούμε αμέσως μέσω αυτής της διαδικασίας την κάλυψη, την αντιστάθμιση του κόστους και των δαπανών διότι αυτά τα στοιχεία δεν έχουν μόνο την πτυχή της αναφοράς και καταχώρησης αυτών των συμβάντων και αντίστροφα πρέπει να ισχύει ότι οι επιχειρήσεις τις σημαντικές για εκείνες, για πληροφορίες πρέπει να μπορούν να τις αντλούν από αυτό τον φορέα η υπηρεσία για τη μέγιστη προθυμία για τη συνεργασία που πρέπει να επιτυγχάνεται πρέπει να δημιουργηθεί ένας περίγυρος εμπιστοσύνης, ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Στα όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 είναι κέρια σημασίας. Η γνωστοποίηση ενός τέτοιου συμβάντος στο επίπεδο ασφάλειας θα μπορούσε να ε, οδηγήσει στην προσέλκυση, στην ε, πρόκληση και άλλων hacker, δηλαδή και άλλων πειρατικών τέτοιων επεμβάσεων. Πρέπει να διασφαλιστεί ένα επίπεδο ασφάλειας Πρέπει να δούμε ότι μπορούν να βλαφθούν με τέτοιο τρόπο οι επιχειρήσει που πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό ο κίνδυνο οπωσδήποτε. Είναι σημαντικό η ασφάλεια δικτύων να είναι πιο αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα να χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για να καλυφθούν τα κενά στην ασφάλεια. Προχώρησα πολύ. Μπορώ να συνοψίσω και να ολοκληρώσω. Έχετε ήδη ξεπεράσει το χρόνο σας. Μετά μπορούμε να φέρουμε κάποια σημεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χρησιμότατη η αρχή. Ξέρουμε τι να δούμε όσον αφορά το άρθρο 14 και το άρθρο 12. Αυτό ήδη το απομνημόνευσα. Ας πάμε στον επόμενο μιλητή. Την παρουσίασα, την κυρία Ράτ. Ε, θα μιλήσει ήδη για τη δουλειά που έκανε και κάνει σαν μέλος ε, κυβερνήσεως ενός, ε, της κυβερνήσεως ενός κράτους μέλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που μιλώ μπροστά σε τέτοιους επιφανείς ε, ακροατές και καλούς συναδέλφους. Πολλοί από αυτοί, πολλοί από αυτούς έχουν ακούσει πολλά για την όλη εξέλιξη του κυβερνοχώρου στην Εστονία και βέβαια βασίζεται στα γεγονότα του 2007. Όμως τις διαφάνειες όσον αφορά τα οργανωτικά στοιχεία και τις οργανωτικές κυβερνητικές δημές του κυβερνοχώρου στην Εστονία θα σας δώσω κάποια στοιχεία εντάχει αλλά έχετε τις διαφάνειες και νομίζω ότι εξηγούνται από μόνες τους. Είναι αυτονόητο το νόημα. Λοιπόν, τι είδαμε. Και αυτή είναι ήδη παλιά διαφάνεια που βλέπετε. Είναι ήδη τριών ετών ο νέο κίνδυνος, η νέα απειλή, το παράδειγμα, το μοντέλο νέας απειλής, είδαμε νέο κίνδυνο, νέα απειλή υπάρχει σε να αναφέρεται λόγω της τεχνολογίας και της εξάρτησής μας από την τεχνολογία. Αν η κοινωνία της Εστονίας δεν ήταν κοινωνία των πληροφοριών, τότε ο αντίκτυπος των επιθέσεων του κυβερνοχώρου του 2007 θα θεωρούνται σαν κάτι ασήμαντο. Όμως, έτσι που θεωρούμε στην νέα στρατηγική του κυβερνοχώρο ή στην ανάπτυξη νέα στρατηγικής, δεν είναι κάτι που είναι αυτόνομο σαν πολιτική. Είναι μια πολιτική, ένα τμήμα πολιτικής που στηρίζει τη στατική για την κοινωνία των πληροφοριών και εξασφαλίζει την καθημερινή μας ζωή, τον τρόπο ζωής μας. Όπως είπε και Άντριο Σφάμπ, δεν αφορά μόνο τα κρίσιμα στοιχεία ε, πληροφοριών του κυβερνοχώρου, αλλά όλη την κοινωνία των πληροφοριών. Πολλοί εδώ στις, στις Βρυξέλλες που θέλουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό ζηλεύουν τους Εστονούς που σε δύο λεπτά ανοίγουν λογαριασμό τραπεζικό και σε πέντε λεπτά μπορούν να συστήσουν μια εταιρεία, άντε δέκα λεπτά. Αλλά ε, αν θέλουμε να εξάγουμε τον τρόπο ζωής μας, τον ηλεκτρονικό τρόπο ζωής, ή αν θέλουμε να δώσουμε διασυνοριακή διάσταση πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, στοιχείο εμπιστοσύνη στην προσπάθεια. Όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτόν τον τομέα, τεχνολογικοί κίνδυνοι, οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι, αυτές είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Πώς βλέπουμε ειναι αυτη ειναι η κατασταση πως βλεπουμε εμεις τις υποδομές και την εξάρτηση, την αλεξάρτηση των τομέων είναι κάτι φέτες στη διαφάνεια. Σε όλη την Ευρώπη είναι παρεμφερής η κατάσταση. βλέπουμε ότι υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις. Και βλέποντας αυτό, είναι μοναδικό το κάθε κάτος μέλος. Έχει διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετική αλληλεξάρτηση των διαφορών τομέων από χώρα σε χώρα διαφέρει. Αυτή είναι η βασική δομή στην Εστονία. Το αναφέρουμε και η στρατηγική μας την πρώτη για τον κυβερνοχώρο. Και πάνω σε αυτή τη βάση που βλέπετε κινούμαστε. Βλέπετε μια δομή οριζοντίου συντονισμού. Υγούνται κυβερνητικά συμβούλια και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και η Διακυβέρνηση. Αυτός ο οριζόντιος συντονισμός, αυτό το σύστημα δεν έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες. Διότι είτε σχετίζεται με την κλίμακα του συστήματος και στο κυβερνοχώρο σε όλο τον κόσμο οι ίδιοι κάθονται γύρω από το τραπέζι όπου και να πας. Ο αντίκτυπος όμως των προβλημάτων στον κυβερνοχώρο είναι κάτι που έχει προτεραιότητα παντού. Ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και τα Υπουργεία θεώρησαν ότι είναι πρόβλημα αυτό. Η Εθνική κατάρτιση εθνικών πολιτικών ξεκινήσαμε το 2007-2008 όταν η φυστάμενη στατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο υπήρχε και η ανάπτυξη πολιτικής θεωρήθηκε βασικό στοιχείο. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Είναι βασικό στοιχείο. Όταν βλέπουμε το θέμα της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστασία κρισίμων πληροφοριών και των σχετικών υποδομών Το τελευταίο δεκάμινο, πριν από δέκα μήνες περίπου, εγώ ήμουν αντίθετη, κάθετα αντίθετη στην επέκταση της ισχύω του άρθρου 13α. Η Εστονία πάντα έλεγε λιγότερες ρυθμίσεις είναι κάτι καλύτερο, είναι περισσότερο. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στις ε, θελοντικές πτυχές ε, διαβίβασης πληροφοριών και ενημέρωσης για τα διάφορα συμβάντα. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. Όμως στην περίπτωση κρισίμων υποδομών πληροφοριακών έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο. Έχουμε προτείνει εθνική νομοθεσία το τελευταίο δεκάμινο να επεκταθεί το 13α σε άλλους τομείς των τηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά την προτινόμενη οδηγία, αυτή είναι πράγματι μια επιτυχία ένα κράτος μέλος έκανε όλα τα βήματα και το σύστημα δουλεύει. Δουλεύει για μα. όμως. Πιο συγκεκριμένα. Βλέποντας το ιστονικό μοντέλο που είναι πολύ εύκαμπτο Υπάρχουν στόχοι που αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών. Κάτι που διαπνέει τη στρατηγική προστασία ιδιωτική ζωή, ταυτότητα, αυτά τα ήπια μέτρα δεν εντάσσονται στη στρατηγική ασφαλείας του κυβερνόχωρου. Πρέπει να το πω αυτό. Διότι δεν έχουμε ακόμα πλήρως αποφασίσει για τον ορισμό του κυβερνοχώρου. Εστιαζόμεθα και επί των κρισίμων στοιχείων. Αστυνόμευση, εσωτερική ασφάλεια, ευαισθητοποίηση. Αλλά όχι απαραίτητα μόνο αυτό. Κοιτάμε τις ομάδες του πληθυσμού που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν είναι η έφηβοι e και άλλα απλά είδη ε, κυβέρνο Στη συνεργασία μας στην αστυνομία εξετάζουμε το ηλικιακό φάσμα 25 με 45 όπου τα ποσοστά εγκλημάτων είναι πιο υψηλά. αυτού του είδους η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών φορέων, αστυνομίας, κυβέρνησης είναι ύψης της σημασίας. Τώρα, αυτό είναι το στονικό μοντέλο που ακολουθεί στενά από κοντά το μοντέλο που προτείνει η οδηγία, κατά πόσο αυτό το μοντέλο μπορεί να αναπαραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε άλλα κράτη-μέλη, εγώ νομίζω ναι, μπορεί να γίνει, αλλά όχι και τα μέσα. Οι στόχοι που προτείνω στην οδηγία είναι σημαντικότατοι. Όμως, κατά πόσο συγκεκριμένοι θεσμοί και φορείς, η χ, χάρη, μια ομάδα έκτακτης ανάγκης ε, για αντιμετώπιση κυβερνοεγκλημάτων ε, πρέπει να κινείται ακριβώς με πανομοιότυπο τρόπο στη χώρα Α και στη χώρα Β. Δεν έχει σημασία τόσο το μέσο που χρησιμοποιείται, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, η ασφάλεια και η προστασία της τεχνολογίας και της κοινωνίας που εξετάζεται την τεχνολογία. Αυτό εξετάζουμε. Εάν ακολουθήσει κανείς αυτή την προσέγγιση, το μοντέλο μας μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Πρέπει να αναλυθεί όμως με κάθε σοβαρότητα από το συγκεκριμένο κατός μέρος που θέλει να το εφαρμόσει. Δηλαδή, ποιες ε, υπηρεσίες είναι κρίσιμες για τη συγκεκριμένη κοινωνία του συγκεκριμένου κράτους. Ο τραπεζικός τομέας στις περισσότερες χώρες υπάρχει ένα στοιχείο ηλεκτρονικό στις τραπεζικές υπηρεσίες. Θεωρούνται κρίσιμες υπηρεσίες συνήθω. Ο ενεργειακός τομέας. Όλοι είμαστε εδώ χάρη στην ηλεκτρική ενέργεια υπό κάποια μορφή. Ποια τμήματα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρισίμου σημασία εκεί εστιαζόμεθα. Πώς παράγεται, ποια είναι τα μέτρα ανάγκης. Αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα και κατά πολύ. Και η κυβερνοασφάλεια πώς να ενταχθεί στα εθνικά προγράμματα ανάγκης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν είναι κάτι διασυνοριακό και πλήττει πάνω από ένα κάτω μέλος το πρόβλημα, τότε οι κανόνες μπορεί να ποικίλουν. Ε, εξετάσαμε με κάθε σοβαρότητα τις διάφορες διαργασίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μαζί με την ΕΝΗΣΑ αλλά όσον αφορά τις εθνικές αντιδράσεις, εθνική κρίση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της κάθε κοινωνίας. Τώρα αν υπάρχει μεγάλη φορά μεταξύ εφαρμογής αυτού του είδους του μοντέλου σε χώρες που είναι πιο προχωρημένες τεχνολογικά ή που εξαρτώνται περισσότερο από την τεχνολογία ή έχουν μείνει πίσω στο χώρο τον ηλεκτρονικό, τον κυβερνοχώρο δύσκολο να πει κανείς ότι έχουν μείνει κάποιες χώρες πίσω Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που διαπιστώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εταίρους Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξή. Οι ασκήσει οι ευρωπαϊκές, της Ευρωπαϊκής Ενώσεω όσον αφορά τον κυβερνοχώρο. Η άσκηση που έγινε το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ επιτυχής. Ε, ενδιαφέρθηκαν πολλά κράτη-μέλη και οργανισμοί, οι υπηρεσιών των κρατών μελών διαφέρθηκαν. Εκεί είδαμε ότι είχαν αυξηθεί οι πάροχοι υπηρεσιών εκθετικά σε αριθμό και δεν μπορείς να κάνεις μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ Εστονίας και κάποια μεταξύ με άλλες χώρες όπου η ασφάλεια του κυβερνοχώρου δεν θεωρεί το πολιτική προτεραιότητα. Θα πρέπει ο κυβερνοχώρος να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι σε μια στρατηγική του κυβερνοχώρου και στα σχέδια δράσης στα συναφή ε, πρέπει να συνυπολογίζει κανείς και το κόστος από τον εθνικό προϋπολογισμό. Και το κόστος για την ασφάλεια δεν δίνει άμεσα αποτελέσματα απαραίτητα, αν κοιτάξει κανείς τα συγκεκριμένα, τους συγκεκριμένους στόχους στην κυβερνοχώρο. Όμως, αν όπως στην Εστονία δει κανείς την ανάπτυξη κοινωνία των πληροφοριών, ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα κέρδη, για τις επιχειρήσεις και τον πληθυσμό και τι αναμένουν να κερδίσουν, τότε οι επενδύσεις αξίζουν. Τώρα πώς αυτό θα οργανωθεί σε άλλες χώρες, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο να εξηγήσει κανείς αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αυτή τη στρατηγική, μεγάλη στρατηγική και προστατεύουμε αυτές τις υποδομές. Γιατί το κόστος αποθαρρύνει. Αλλά τώρα πλέον αυτό γίνεται συνηθισμένο. Οι δομές πρέπει να αλλάξουν. Ο, ο πανεπιστημιακός ερευνητής μέσα μου λέει ότι ο Αριστοτέλης κατέληξε σε έξι θεσ, θεσμούς για το κράτος. Μετά τις τεχνολογικές επαναστάσεις πιο πολλοί ε, θεσμοί έχουν δημιουργηθεί ε, οικονομία, μεταφορέ κλπ. Εξελίξεις στου διάφορου τομείς. Και αυτή είναι άλλη μια τεχνολογική επανάσταση. Ίσως χρειαστεί 10-15 χρόνια, αλλά τελικά, τελικά τα πράγματα αλλάζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για, αυτά που μας είπατε, όπως επίσης και για τη φιλοσοφία που μας αναπτύξατε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά ε, σε σχέση με τις ε, δυνατότητες που δίνει αυτή ε, η πρόταση. Ο Ολιβιέ Μπουργκεστάικ ε, αναμένουμε αγωνίως να ακούσουμε τι θα μας πει. 15 λεπτά το πολύ. Αλλά αν μας τα πείτε και σε λιγότερο χρονικό διάστημα θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ε, εγνωμοσύνη μου που ε, με καλέσατε εδώ εκ μέρους ε, της Europol. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, είναι πολύ τομεακή υπό διάφορες οπτικές γωνίες προσπαθεί να ε, αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επίσης ε, βλέπει περισσότερο προς το μέλλον. Οι επιχειρήσεις μας, ε, οι υποδομές δεν είναι υπερφορτωμένες ακόμα και μπορούν να λειτουργήσουν σχετικώς καλά. Αλλά αυτό για την ώρα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον και το να ε, προβλέπουμε ε, διάφορες καταστάσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας. Αυτά ε, που είδαμε σε σχέση με το κείμενο είναι απλώς κάποιοι πρώτοι άμεσα επιτεύξιμοι στόχοι, ό,τι έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα και αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη την αυξανόμενη εξάρτησή μας από το διαδίκτυο στις κρίσιμες υποδομές μας και στις επιχειρήσεις μας, πρέπει να είμαστε να λάβουμε τα σωστά μέτρα. Τώρα, τι χρειάζεται για να κάνει κανείς ένα έγκλημα μέσω ίντερνετ. Δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα. Τα εργαλεία ε, βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικό ε, στο ίντερνετ για να διαπράξει ένα έγκλημα. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τα σωστά μέτρα. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ε, ευελιξία για να μπορούμε να για να μπορούμε να, να, όταν συμβαίνει κάτι να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και για λόγους πρόληψης και για λόγους ε, διακοπής ορισμένων δραστηριοτήτων γιατί το γεγονός ότι η πρόταση αφορά ήδη ε, το, το γεγονός ότι ε, η κρίσιμη υποδομή λαμβάνεται υπόψη είναι νομίζω πολύ καλό. Η ανταλλαγή πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις εκ των προτέρων το, όσο το δυνατόν ε, περισσότερο, όπως επίσης επιβολή του νόμου μόνο στις περιπτώσεις όταν υπάρχει ε, λόγος να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να είναι επί εγκληματικής φύσεως μια δραστηριότητα, νομίζω ότι καθιστά την πρόταση ισορροπημένη. Όσον αφορά τώρα το, την άποψή μας ε, ως Ευρωπαϊκού ε, Κέντρου ε, πρόληψης του εγκλήματος μπορούμε να υποστηρίξουμε ορισμένα στοιχεία της πρότασης ως τρόπο να καταστήσουμε την Ευρώπη ασφαλέστερη. Όταν ε, μιλούμε για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ε, εγκληματικής φύσεως, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να ε, τα λάβουμε υπόψη και έχουμε το, τα δίκτυα και έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ε, γρήγοροι στην αντιμετώπιση μας και ε, να ε, επιλύσουμε τα προβλήματα όσο το δυνατόν συντομότερο. Όσον αφορά τώρα τις προκλήσεις που έχουμε λόγω των διαφορετικών νομοθεσιών, έχουμε χρόνια εμπειρίας και έχουμε ένα δίκτυο εσωτερικό που μπορεί να μας βοηθήσει σε γρήγορη ανταλλαγή απόψε πληροφοριών και συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν ε, οι διάφορες πηγές αυτής της πρότασης μας βρίσκουν ε, σύμφωνους. Όπω είπα και προηγουμένω, μπορώ να πιστέψω βέβαια ότι για κάποιε από τι επιχειρήσει είναι λίγο πρόημο να καταλάβουν από τώρα ε, το λόγο ύπαρξη αυτή τη πρόταση, αλλά θα το καταλάβουν όταν θα είναι θύματα μια επίθεση. Από απόψε ω επιβολή του νόμου Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση αυτή. Βεβαίως θα βοηθήσουμε και εσά αλλά και τι επιχειρήσει στην προσπάθειά σας να ε, το ε, προωθήσετε. Ευχαριστώ. Well, thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Μετά θα πάμε στο επόμενο πάνελ και θα έχουμε συζήτηση και μετά. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο? Αντρέας Φάμπ, μήπω έχει ερωτήσει να θέσει. και αν θέλει κάποιο, κάποιος άλλος συνάδελφος ε, να θέσει ερωτήματα, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προς την κυρία Κίζο μία ερώτηση θα είχα, αλλά με την ανταλλαγή νομίζω στο δεύτερο γύρο του πάνελ μπορεί καλύτερα αυτό να ενταχθεί στη συνέχεια. Γι' αυτό μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Εσθονίας, μιας χώρας που έπρεπε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους επιθέσεις ήδη. Είπατε ότι ο ορισμός ε, της κέρια κριτικής υποδομής στο τέλος τέλος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και από χώρα σε χώρα είναι διαφορετικό ζήτημα. Θα ήθελα όμως εδώ να σας παρακαλέσω παρόλα αυτά την προσωπική σας άποψη να μου πείτε. Τον ορισμό αυτόν πώς τον εκτιμάτε, αυτόν που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον μη εξατλητικό κατάλογο, non-exhaustive list. Κυρίως θα με ενδιαφέρει η δική σας εκτίμηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τις ε, κυβερνοϊπηρεσίες σε σχέση με αυτά τα δίκτυα. Στην Εστονία αυτά διαδραμάτισαν κάποτε κάποιο ρόλο. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Ίσως κάτι θα μπορούσατε να μας πείτε σχετικά. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και μετά θα δώσω τη δυνατότητα σε κάθε προσκεκλημένο να απαντήσει. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας. Συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερους συναδέλφους παρόντες. Η ποιότητα της παρουσίασής σας είναι εξαιρετική και θα ήθελα να απευθυνθώ ε, προς την εστονή προσκεκλημένη μας. Ε, μιλήσατε για τους ορισμούς, το είπε μόλις και ο Ανδρέας. Ε, καλύτερα να έχουμε αποτελέσματα, αλλά όχι τόσο όρους, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Ε, σωστό είναι αυτό, αλλά είχατε αυτή την εμπειρία μια απειλή στο σύστημά σα, ένα σύστημα που θα θέλαμε να έχουμε εμεί στι χώρε ε, μα. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε με περισσότερε λεπτομέρειε. Τα ακούσαμε βέβαια, το διαβάσαμε σε εφημερίδε, αλλά εσεί είχατε άμεση εμπειρία. Τι μάθατε από αυτό. Μιλήσατε λιγάκι γι' αυτό, αλλά τώρα ε, που τι θα κάνατε διαφορετικό και επίσης για τις συζητήσεις ε, για την προστασία των ε, δεδομένων. Όλες αυτές τις συζητήσεις που τις είχαμε πιο σύντομα, πιο πρόσφατα σε σχέση με ε, την συζήτηση που κάνουμε σήμερα. η ισορροπία του ιδιωτικού βίου αλλά και της ασφάλειας ήταν κάτι που σας απασχόλησε, ήταν τμήμα των προκλήσεων που είχατε να αντιμετωπίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ως Πρόεδρος ε, θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα ε, προς όλους εσάς ε, μου άρεσε αυτό που είπε η κυρία Κίσουφ ε, σε σχέση με τις βασικές πτυχές της συνεργασίας και πώς αυτό ήταν μια σημαντική επιχειρηματική στρατηγική για τις ε, ε, εταιρείε. Κάτι άλλο όμως το οποίο προκύπτει όμως και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπε και η κυρία Ράουντ για την αλλαγή της προσέγγισης. Είναι μη ρεαλιστικό να επιβάλλει κανείς τη συνεργασία, γιατί η συνεργασία θεωρείται ότι εξορισμού είναι κάτι το εθελοντικό. Μήπως θα, μπορούσε, μήπως θα είναι αντιπαραγωγικό το να υποχρεώνει κάποιους να συνεργαστούν, ε, κάποιους να, τους υπόλοιπους να συνεργαστούν. Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα προκύψει και στις δικές μας συζητήσεις ως πρόβλημα. Τι είδους, ε, τέτοιου είδους ε, κίνητρα μπορούμε να δώσουμε, για παράδειγμα βέλτιστες πρακτικές, ε, ε, για να ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο. Αν, Ανδρέας, θέλεις να πεις κάτι ακόμη? Πρόεδρε, μια ερώτηση ξέχασα. Ο εκπρόσωπος ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας καταρχήν διατύπωσε κάποια ερωτήματα. Εμένα ως αντερώτημα θα με ενδιέφερε Μπορείτε να δώσετε μια σύντομη περίληψη, μια σύντομη σύνοψη. Ποιε συγκεκριμένε τέτοιε ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ ε, του δικού σας οργάνου και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων γίνεται για την κυβερνοασφάλεια. Κατά κάποιο τρόπο βρίσκεστε, βρίσκεστε εσείς εμπλεκόμενος σε αυτό το πεδίο. Τι απορρέει από τις επαφές σας με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να παράγουν τις περισσότερες πληροφορίες. Αυτό θα με ενδιαφέρει σε σχέση με αυτά που είπε και ο Πρόεδρος. Αυτή η αγορά διοργανώνεται επί επί εθελούσιας βάσης, έτσι δεν είναι. Okay. Uh, well... Πολλές ερωτήσεις προς την κυρία Ράουντ. Ε, να ε, σας ε, δώσω το λόγο εσάς πρώτα, μετά η κυρία Χίσουφ και μετά ο κύριος Πουρτεστάικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, καταρχάς όσον αφορά του ορισμούς ε, του κυβερνοχώρου και τη ε, σχέση των ορισμών με τους τρόπους και τα, τα μέσα και τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο ευχαρίστω θα είχα συζητήσει πριν από τρει μήνε, πριν από την αναθεώρηση τη κυβερνοστρατηγική τη Εστονία. Όμω δυστυχώ ε, εγώ στι ομάδε εργασία μου το έθεσα αυτό το θέμα και δεν έχω ιδέα προ τα που οδεύουμε. Το θέμα είναι σήμερα ότι έχουμε πάρα πολύ προχωρήσει από αυτό το υπολογιστή ε, δίκτυο ε, πλέον. Το 2007-2008 καταλαβαίναμε ότι υπήρχαν τέλος πάντων κίνδυνοι, απειλές... Ε, όμως σήμερα η απειλή αφορά το κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία στην όλη διαδικασία δεν αφορούν μόνο του υπολογιστέ, δηλαδή. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να πω δυστυχώς το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε οποιοδήποτε άλλος ε, συμμετέχει στην προετοιμασία της οδηγίας σε έξι μήνες θα μπορέσω να σας πω για το 2007 και την εμπειρία μας ε, από την απειλή που είχαμε και το τι μάθαμε, δεν ήταν τόσο οι τεχνολογικές επιθέσεις, ε, γιατί ε, η άρνη, η, επιθέσεις σε υπηρεσίες ήταν κάτι που το γνωρίζαμε από πριν. Το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκαν ε, εξεγέρσεις, ε, υπήρχαν κοινωνικά προβλήματα, ε, υπήρξε μια ολόκληρη πολιτική ιστορία γύρω από αυτό και οι επιθέσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ως πολιτική δήλωση. Χρησιμοποιήθηκαν τα κοινωνικά μίντια, χρησιμοποιήθηκε ο κυβερνοχώρος που είναι προσβάσιμος από, από τα κινητά τηλέφωνα. Υπήρξαν και αντίπεινα. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε Επιτροπή, σε ε, ε, διάφορα άλλα μέσα. Το mass messaging, τα πολλά μηνύματα. Ε, η εξάρτηση από την τεχνολογία και σε πολιτικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παίρνει κανείς πολύ σοβαρά. Από την άλλη με ρωτήσατε επίσης για την ε, προστασία των δεδομένων, τον ιδιωτικό βίο και ε, κατά πόσο έπρεπε να ασχοληθούμε και με αυτό. Η στρατηγική μας δεν επικεντρώνεται ε, σε ζητήματα ιδιωτικού βίου. Στην πράξη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα από την κοινωνία, από τον χρήστη όλων αυτών των, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και όλων των σχετικών αυτών μέσων, είτε είναι η φύση των στονών, είτε είναι το γεγονός ε, ότι μέχρι τώρα ηλεκτρονικές υπηρεσίες ε, ε, μέσω του X-Road, δηλαδή της πλατφόρμας από την οποία περνούν τα πάντα, δεν έχει προσβληθεί ε, ακόμα. Αυτό ε, ισχύει τα τελευταία δέκα χρόνια, οπότε υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και στην Εστονία. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες υπήρχαν συζητήσεις ε, για, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά πόσο κάποια στοιχεία της δικής σου ταυτότητας, όπως για παράδειγμα η φωτογραφία σου ή υπόλοιπες, ε, τα υπόλοιπα στοιχεία της ταυτότητάς σου ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην Εστονία δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Θεωρήθηκαν αυτά τα πράγματα δεδομένα. Για τη γενική ερώτηση που κάνατε εσείς κύριε Πρόεδρε σε σχέση με την εμπιστοσύνη κατά πόσο μπορεί κανείς πραγματικά να ρυθμίσει την εμπιστοσύνη. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήμασταν τυχεροί στην Εστονία από αυτή την άποψη λόγω των κυβερνοπιθέσεων, γιατί συνεργάστηκε ο ιδιωτικό τομέα και παρέμεινε ε, ενωμένο. Οπότε έχουμε μια ε, ε, ρυθμιστική υποδομή και τώρα υπάρχει το ΣΥΖΟ, διάφορα άλλα δίκτυα ε, μετά από το 2007, μετά ε, τη χρονική στιγμή που ε, άρχισαν να δουλεύουν μαζί, συνέχισαν να συνεργάζονται. Οπότε Έτσι μόνο δουλεύει η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών. Όταν ο ιδιωτικό τομέα θα πάει στην κυβέρνηση και θα πει πρέπει οπωσδήποτε να επισημοποιήσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πραγματικά είναι ο κυριότερος παράγοντας της συνεργασία, της ε, εθελοντικής συνεργασίας που είναι η εμπιστοσύνη ο πιο, αποτέλεσμα, ο πιο ο κυριότερος παράγον. Και τώρα φανταστείτε ότι τα ιδιωτικά σας προβλήματα θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να τα καταχωρείτε κάπου. Κανένας δεν θέλει να το κάνει αυτό ευχάριστα. Κοστίζει και χρήματα, είναι δαπανηρό να καταχωρείτε αυτό. Υπάρχουν και πολλές επιφυλάξεις να γίνεται αυτό. Θα πρέπει όμως να δούμε τα κίνητρα. Τα κίνητρα μπορούν να δοθούν με τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τις επιχειρήσεις. Αν τραβάμε όλοι ένα σκηνή προς μια κοινή κατεύθυνση και δουλεύουμε όλοι από κοινού για την ε, αύξηση της ασφάλειας ε, στο δίκτυο από πλευράς ασφάλειας με σκόπιμες ε, στοχοθετημένες εξειδικευμένες πληροφορίες θα συνεργάζονται οι εταιρείες όταν θα υπάρχει δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων ή όταν θα υπάρχει δυνατότητα μιας δεξαμενής που θα δίνει προτάσεις για την επίλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται απλά και μόνο με τη δημοσιοποίηση μιας, ότι σε μια επιχείρηση έγινε τούτο ή το άλλο και αυτό ήταν σημαντικό. Αυτό δεν έχει το σημαντικότερο ρόλο. Το σημαντικό θέμα είναι τα θέματα ασφάλειας που πρέπει να αποκαλύπτονται. Θα έχει και μεγάλο αποτέλεσμα για το ήπιο, για το λογισμικό, software και hardware, ότι θα μπορούσε κανείς ε, να έρθει στην ιδέα δημοσιοποίησης κάποιων στοιχείων η αποκάλυψη και δημοσιοποίηση είναι κάτι πιο αποτελεσματικό για την ασφάλεια από ότι η έγερση κάποιων κατηγοριών ή απλά η καταχώρηση κάποιου συμβάντος. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία με κάποιον επειδή απορρέει κάποια πρόσθετη αξία από, αυτό, από αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Στην Europol Είχαμε πολλέ ρυθμίσει όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και σοβαρή είναι η υποπτία. Διότι αυτό βοηθά διότι ελέγχουμε φοβερά την επεξεργασία των δεδομένων και δημιουργείται εμπιστοσύνη μεταξύ ημών ε, και με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τους ιδιωτικούς ε, εταίρους. Μπορεί να μας δώσουν στρατηγικές πληροφορίες οι ιδιωτικοί εταίροι, μη προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα μπορούν μόνο με εθνικών αρχών να τα κοινοποιήσουν και των εθνικών μονάδων και τότε καταφθάνουν σε εμά. Η Εθνική Αρχή έχει την ευθύνη γι' αυτό. Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε σε ιδιωτικούς φορείς. Αλλά πρόσφατα είδαμε όσον αφορά το κυβερνοέγκλημα ότι κάποιοι ιδιωτικοί φορείς είναι πρόθυμοι να δώσουν πληροφορίες όσον αφορά τις, πληρο... Ε, απειλές που αντιμετώπισαν ώστε να ενημερωθούν και άλλοι και να προειδοποιηθούν κι άλλοι. και από διάφορε εταιρείε που φτιάχνουν προϊόντα κατά των ιών ε, λαμβάνουμε έγκαιρε προειδοποίησει, από τις εταιρείε που φτιάχνουν αντιβάρου. για να προλάβουμε την μόλυνση και μπορούμε να ενημερώνουμε και κάποιους οι οποίοι μπορεί να απειληθούν από τέτοιου Ιου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ας πάμε στον επόμενο γύρο και αν οι ομιλητές τηρήσουν το δεκάλεπτο θα είμαι ευτυχής, διότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο διάλογο. Να πω κάτι που ήθελα να πω πριν και στο συγγνώμη. Τον κύριο Ζέπε Αλμόντι θα καλωσορίσω και τους συναδέλφους από την DG Connect που ήταν υπεύθυνοι για αυτή την πρόταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε και από αυτόν συντομία κάποια σχόλια, να δούμε πώς θα πάει. Επόμενο. Επόμενος κύκλος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή αντίληψη για το κυβέρνο έγκλημα, τις επιθέσεις, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καινοτοπία και να μεγιστοποιήσουμε τον, τον οικονομικό, τις οικονομικές συνέπειες αυτής της πρότασης. Καλωσορίζω και συγκεκριμένου εμπειρογνώμονε που έχουν ξανάρθει εδώ, στη θητεία μου τουλάχιστον. Ο κύριο Σάμιουλσεν είναι στο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Δικτύων, ΕΝΙΣΑ, Είχα επεξεργαστεί στην πρώτη μου θητεία στο Κοινοβούλιο τη χάρτα για αυτόν τον οργανισμό, εδώ και καιρό. Ήταν και πρόεδρος τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου για το πακέτο τηλεπικοινωνίων όταν κάναμε τη μεταρρύθμιση το 2009. Εκείνοι που συνεργαστήκατε μαζί με από αυτού θα τον ξέρετε. Ε, από την άλλη πλευρά των πραγματεύσεων του υποθετικού τραπεζιού, Ματ Νίλσεν, ε, που έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη τεχνολογίας ήταν επικεφαλής για την έξον για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και εκπροσωπεί και την υπηρεσία του Ινστιτούτου έτσι για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχει συμβάλει και αυτός πολλές φορές συνεδριάσεις και κάποιος που ήρθε για πρώτη φορά και ελπίζω όχι τελευταία, Φλόριαν Γούλφερ από το Κρέος Computer Club που είναι υπεύθυνο, είναι σύμβουλος για την τεχνολογία των πληροφοριών και ξέρει τις αδυναμίες των υποδομών και μπορεί να μας δώσει μια οπτική γωνία για τι πρέπει να κάνουμε. Και τέλος καλωσορίζω το Will Sample από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και το κέντρο για την αντιμετώπιση των απειλών. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τις υποδομές. Θα δώσουμε στον καθένα ένα μερίδιο, δεκάλεπτο, και ελπίζω να κρατήσει το δεκάλεπτο. Ο κύριος Σάμιλσον λοιπόν είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Μάλκον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ Μάλκον που μας καλέσατε σήμερα για να μιλήσουμε. Είμαι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΗΣΑ αλλά είμαι και Σουηδός δημόσιος υπάλληλο που επεξεργάζεται το θέμα, αλλά επικεφαλής είναι ο Ανδρέας Ντόλκης του Υπουργείου Αμήνης, γι' αυτό εμφανίζεται στη διαφάνεια. Και μπορείτε να έθετε σε επαφή μέσω των στοιχείων που σας δίνουμε με τα ονόματα που βλέπετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ σε όλα τα καλά που μπορεί να κάνει η πληροφορική για μας και πόσο σημαντική είναι. Αυτό, αυτή η διαφάνεια επενθυμίζει βέβαια ότι το σύστημα της πληροφορικής πρέπει να δουλεύει όσο ε, θέλαμε. Ξεκινάμε λέγοντας ότι η Σουηδία θέλει ε, υψηλό επίπεδο ασφαλείας των δικτύων πληροφοριών στην Ευρώπη. Είναι καλό για την κοινότητα, για τα μέλη, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση για να πετύχει ακριβώς αυτό το στόχο και κυρίως ε, όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής του του η Σουηδία τονίζει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει διαφορετικές λύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε εκτενώς από τους προλαλήσαντες. Δεν μπορούμε να βρούμε μια γενική λύση. Αυτό που παρουσιάζω είναι η βασική μας αντίδραση. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Μου είπα να αναλύσω την άποψη της ε, Σουηδίας για τα θέματα της επικουρικότητας που έθεσε το Σουηδικό Κοινοβούλιο. βασίζεται σε ένα πρώτο προκατακτικό υπόμνημα που του στείλαμε και στέλνουμε υπομνήματα για άλλε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την ίδια άποψη όπω το κοινοβούλιο μα. Ίσως ε, να θεωρείτε ότι έχω μία τάση αντιπαράθεση με αυτά θα πω, αλλά ε, ε, οπότε γίνεται πιο δύσκολη η κατάσταση γιατί πρέπει να τα περιγράψω όλα πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έλλειψη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα οδηγούσε σε δράση κρατών μελών μεμονωμένα. Και δεν θα λαμβάνεται υπόψη ελεξάρτηση των διαφόρων δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ήδη λαμβάνει η χώρα συντονισμό. Τα ανέφεραν και άλλοι προλαλήσαντε. Βασίζεται σε ευελιξία και εμπιστοσύνη. Ακούσαμε επανειλημμένα ότι η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να επιβληθεί. Δεύτερον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφορε νομοθεσίε των κρατών μελών για το σύστημα αυτό ασφαλεία για, ε, για την πληροφορική εμποδίζει τι διάφορε επιχειρήσει που θέλουν να κινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασυνοριακά και υποχρέσει ε, που επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργούν ισότιμους όρους για όλους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εταιριών του τομέα που λειτουργούν σε πολλά κράτη-μέλη και σε όλη την Ένωση παρά τις διαφορές της νομοθετικές και παρά τα επίπεδα ασφαλείας και δεν βλέπουν να υπάρχουν σαφή στοιχεία ατελειών της αγοράς τουλάχιστον από την αξιολόγηση συνεπειών που έχει δοθεί. Και τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται μεμονωμένα ε, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρας και ανάλογα με το κόστος και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται και όχι με μια ενιαία προσέγγιση. Για την επικουρικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μια εκούσια εφαρμογή οδήγησε σε μια συνεργασία της μειοψηφίας των κρατών μελών που έχουν μεγάλες δυνατότητες ε, προστασίας. Δεν νομίζουμε ότι αυτό, αυτή η δήλωση ε, ευσταθεί όσον αφορά τη δημιουργία λεπτομερούς νομοθετικής κάλυψης επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως η, χαμηλή, η μικρή δυνατότητα δεν είναι ε, βασική αιτία για την έλλειψη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, περισσότερο εμπιστοσύνη. Με βάση άλλου παραμέτρου. Είναι και θέματα πάπτονται εθνική ασφαλεία. Βασικό παράγων που δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πιστεύουμε όμω ότι είναι σημαντικό να ανεβεί το ελάχιστο επίπεδο προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάρτιση συντονισμού συστάσεων ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ελευθόρων λεπτομεριακών διατάξεων. Χτες πήρα στοιχεία από τη δικό μας φορέα που έδειξε κατάλογο χωρών που έχει το μικρότερο αριθμό ε, μολυσμένων ιών. Εμείς είμαστε υπαριθμόν 4 στον κατάλογο. Και το καταφέραμε αυτό χωρίς να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία για τους τελικούς χρήστες, και τις εταιρείε σε μεγάλο βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τονώσει την αποτελεσματικότητα εθνικών στρατηγικών. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια χώρα που αγνοεί τις απειλές. Αλλά έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την νομοθεσία, πόσο περιοριστική πρέπει να είναι. Να θέλουμε να έχουμε μια γενική στρατηγική είναι ένα πράγμα. Το τι ακριβώς θα περιέχει η στρατηγική είναι κάτι διαφορετικό. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι τα μέτρα της ασφαλείας των δικτύων που λαμβάνονται από κυβερνήσεις πρέπει να είναι συντονισμένα για να αρχιστοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν τα επεισόδια στον τομέα της ασφαλείας. Αν υπάρξει επεισόδιο, συμβάν, πρέπει πρώτα ακαρία να αντιμετωπιστεί το συμβάν. Και τότε κάποιος να αποφασίσει επιτόπου πότε και με ποιον έρχεται σε συνεννόηση και συντονισμό. Το είδαμε από ασκήσει που κάναμε μαζί με άλλα κάτι μέλη ότι πολύ συχνά είναι καλύτερο κάποιο που έχει πληγεί αλλά λιγότερο να συντονίζει και να ενημερώνει τους άλλους. Ανταπόκριση συντονισμένη σε κάθε συμβάν ίσως να είναι κάτι πολύ αρνητικό. Πάμε στην αναλογικότητα. Η αρχή της αναλογικότητας απαιτείται από τα κράτη-μέλη στην πρόταση να κάνουν πράγματα όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο για να υπάρχει ε, επαρκή ετοιμότητα και να υπάρχει και εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συνεργασία. Σαν να παπαγαλίζω, αλλά θα το πω, αυτή η συνεργασία χρειάζεται υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη, κάτι που δεν επιβάλλεται. Αυτό πιστεύει η Σουηδία. Και η ΕΝΙΣΑ, ο φορέα για την ασφάλεια του δικτύου, ήδη λαμβάνει μέτρα για ευαισθητοποίηση για να αυξήσει την ασφάλεια των δικτύων και τι δυνατότητε αμήνη στην Ευρώπη. Η ΕΝΙΣΑ διευκολύνει και πολλαπλασιάζει τις προσπάθειες αντίδρασης, την δημιουργία, την, την απόκτηση γνώσεων, προσόντων κλπ. Για την αναλογικότητα, διατείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων αφορά μόνο κρίσιμους ε, φορείς και όλα τα άλλα εξαρτώνται από το κόστος και το κίνδυνο. και πρέπει να δίνονται αναφορές μόνο για σημαντικά συμβάντα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι κρίσιμη φορείς είναι κάτι πολύ αόριστο στην πρόταση και τα μέτρα ασφαλείας και αναφορά συμβάντων είναι κάτι που πολύ συχνά δεν αντιστοιχεί ούτε στους κινδύνους ούτε στο κόστος που συνεπάγονται οι κίνδυνοι. Και πρέπει να υπάρχει γενική εξαίρεση για την υποβολή αναφορών και εκθέσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας όπως αμυντικά ζητήματα. και άλλα θέματα που, και προβλήματα που βλέπουμε. Ένα αφορά την βάση, την ενιαία αγορά. Ήδη τα ανέφερα ακροθυγός. Οι πτυχές ανταγωνισμού και ισότιμες συνθήκες για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό δεν είναι κάτι σχετικό. Και η προτινόμενη νομική βάση για την ενιαία αγορά με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται πολύ σχετική. Υπάρχουν πιο κατάλληλες νομικές βάσεις συνθήκη όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας που αφορούν περισσότερο την ασφάλεια και όχι τόσο πολύ τα θέματα ανταγωνισμού και ενιαίας αγοράς. Όμως, περαιτέρω διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς, ελπίζουμε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για μελλοντικές προοπτικές αγοράς και τις σημερινές συνθήκες αγοράς. Να τονίσω και την αρχή της ευθύνης. Όλοι, όλοι οι κάτοχοι συστήματος πληροφορικής πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία. Οι κυβερνητικές αρχές δεν πρέπει να δημιουργούν την εικόνα ότι μπορούμε να δώσουμε μια σπίδα που αποφεύγει τους κινδύνους, ούτε και μια εικόνα ότι πάντα θα υπάρχει μια ομάδα που θα σώζει το κοινό από συμβάντα. Αλλιώς δεν, αν τα κάνουμε αυτά δεν θα επομιστούν όλοι τις ευθύνες και δεν θα δημιουργηθούν, δεν θα προστατεύονται παρκώς οι υποδομές του διαδικτύου. Όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές, βασική προτεραιότητα είναι ότι η οδηγία δεν πρέπει να υποχρεώνεται κάτι μέλη να αλλάξουν τις δομές που έχουν και τις ευθύνες που υπάρχουν και κατανεμηθεί μεταξύ εθνικών φορέων αποφασίζοντας επί μίας και μοναδικής αρμόδιας αρχής ε, για την ΕΝΙΣΑ να σας πω κάποια πράγματα εφόσον είμαι εδώ σαν πρόεδρος αυτού του οργανισμού είναι το κέντρο αριστείας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι διαθέσιμο σε όλους και το σέβονται όλοι κάναμε συστάσεις Έχουμε προχωρήσει πολύ. Έχουμε βρει απαντήσεις για προλήψεις κατά των επεισοδίων συμβάντων κινδύνων. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ χωρών, μεταξύ του επιχειρησιακού προσωπικού. Χρειάζεται συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, διότι και η γνώση του είναι σημαντική. Διότι και βασικά αυτοί κατασκευάζουν και υπερασπίζονται τα συστήματα πληροφορικής επί των οποίων εξαρτώμεθα η ΕΝΗΣΑ, δίνει βάση για συνεργασία και διευκολύνει τις προσπάθειες. Εφαρμόζοντας την οδηγία, θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να αφήσουμε την ενίσα να κάνει τα δέοντα στα πλαίσια της νέας εντολής που θα ισχύει από αύριο και το επιχειρησιακό προσωπικό που θα πάει στην Αθήνα με όλα αυτά εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να πετύχουμε το σκοπό και να εκπληρώσουμε το καθήκον που μας ανετέθη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ χειροπιαστές συγκεκριμένες απόψεις. Θα είναι στα φυλάκια, μας φαντάζομαι η τεκμηριωμένη αυτή τοποθέτησή σας. Δεν έχει ίσως συζητηθεί, αλλά όντας παλέμαχος σε σχέση με τις αρχικές συζητήσεις στην Ενίσα, είχε περισσότερες φιλοδοξίες και στόχους αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τους όρους το να πλησιάσουμε, προσεγγίσουμε περισσότερο αυτά τα οποία προτείνονται τώρα όσον αφορά και τα κράτη-μέλη έχει ήδη, α το πω έτσι, δημιουργήσει ευδιάκριτα τις τοποθετήσεις της ε, η ΕΝΗΣΑ για την βέλτιστη συμμετοχή και διάχυση πληροφοριών. Και τούτων λεχθέντων να προχωρήσουμε στη συνέχεια να ακούσουμε από τον κύριο Νίλσον από την ΕΤΣΙ τι γίνεται σε σχέση με, με, τις μελλοντικέ ε, κατευθύνσεις όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές σε αυτό το πολύ σημαντικό πεδίο. Έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήδη αναφέρθηκε πιο πριν. Προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές. Πολύ σημαντικά εργαλεία ως μέσα για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση σε μια ευρύτερη αγορά. Επίσης είναι, χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερο βαθμό στο πλαίσιο αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας. Θα κάνω λόγο λοιπόν για το πώς ε, από πλευράς έτσι και τι γίνεται και με τις προδιαγραφές όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές που αναπτύσσονται για τις βέλτιστες προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας στο χώρο αυτό. Έτσι, Παράγουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία σε σχέση με την πληροφορική και το διαδίκτυο και αναγνωρίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΦΤΑ, αναγνωρίζεται αυτό, παράγουμε αυτά, αυτές τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και το, τις προδιαγραφές GSM που είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Έχει 750 μέλη παγκόσμια. Είναι μια παγκοσμιοποιημένη οργάνωση. 30.000 δημοσιεύσεις έχουν ήδη γίνει που είναι ελεύθερα προσπελάσιμες στο, στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά. Στον τομέα της ε, κυβερνοασφάλειας στο δίκτυο Ήδη όσον αφορά τις εργασίες μας εντάσσεται αυτή η πτυχή. Τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αναπτύσσονται μέσω της ομάδας εργασίας έτσι που τώρα χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στο GSM και στην τελευταία γενεά, της τέταρτη γενεά των τηλεπικοινωνιών και σε άλλα μέσα. Η αντιμετώπιση λοιπόν προδιαγραφών ασφάλειας για το δίκτυο επόμενης γενεάς, δηλαδή τα εξυγχρονισμένα δίκτυα για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και παρόμοιων τεχνικών όπως Do Light Radio και άλλες σύγχρονες πρακτικές όπου να ε, δημιουργείται ένα πλαίσιο ασφάλειας καθορίζοντας τι είναι εκείνο που και με ποια αιτήματα θα μπορούσαν να διαβιβάζονται ε, δεδομένα από τα δίκτυα προς τις αστυνομικές αρχές και άλλους φορείς. Μόνο συγκεκριμένα εξειδικευμένα στοιχεία και μετά από μια τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών όσον αφορά προθεσμίες και διαδικασίες, ε, υπογραφές, smart codes, ε, μηχανή προς μηχανή, συσκευή προς συσκευή, ευφυείς τηλεπικοινωνίες. Εμπλεκόμαστε σε πολύ προηγμένες τεχνολογίες όσον αφορά τις προδιαγραφές ε, που σχετίζονται με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την κωδικοποίηση και την αποκρυπτογράφηση και κρυπτογράφηση με τους δείκτες ασφάλειας στην πληροφορική κτλ ένα τμήμα αυτών των δραστηριοτήτων ε, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων και ε, προδιαγραφών που εκπονούνται για την ε, κινητή τηλεφωνία και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Συμμετέχουμε και στον συντονισμό, ομάδα συντονισμού για την ασφάλεια που είναι κάτι ε, με ευρύτερη εμβέλεια. Επικεντρωνόμαστε σε σχέση με τις σωστές προδιαγραφές που πρέπει να εξευρεθούν και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των κέριων υποδομών. Εξετάζουμε επίσης το τι τεκταίνεται όσον αφορά ε, τους ε, υπολογιστές μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερης δικτύωσης υπολογιστών στο cloud computing. Επίσης εξετάζουμε σε συστήματα διαβίβασης ιατρικών δεδομένων, ε, κινητών ε, τέτοιων ε, δυνατοτήτων και συσκευών, δηλαδή ιδιαίτερα ισχυρών και αποδοτικών ηλεκτρονικών εγκεφάλων, machine to machine, κάνοντας λόγο για το, ε, αυτά τα δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή σε ελεγχόμενο χρόνο, σε πραγματικό χρόνο ε, ελέγχοντας και τα δίκτυα ε, διαβίβασης, ηλεκτρικά δίκτυα κτλ. Πράγματα πολύ σημαντικά για την ασφάλεια. Πτυχές που συσχετίζονται με την ταυτοποίηση ή τον εντοπισμό και άλλες τεχνικές ασφάλειας όπως ηλεκτρονικές ταυτότητες και δημόσιες τέτοιες υποδομές. Επίσης ε, για την ανταλλαγή δεδομένων, πώς θα έπρεπε να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και hm, ταυτοποίηση ψηφιακών στοιχείων, πώς θα μπορούσαν σε κάποιους τομείς δηλαδή να υπάρξουν δράσεις ε, μέγιστης αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι η γενική εικόνα ο ε, σκηνικό α, των όσων γίνονται σήμερα. Έχουμε κάποιες προδιαγραφές πιο τεχνικού χαρακτήρα για τη λειτουργικότητα της ασφάλειας κλειδάριθμους, αλγόριθμους για την αποκρυπτογράφηση και κρυπτογράφηση. Αυτό είναι μια δραστηριότητα πυρήνα στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας ε, που βρίσκεται ως αιχμή του δόρατος στην βελτίωση της ε, διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας. Και φυσικά το έτσι Επίσης έχουμε και, είμαστε και εταίρος και ομόλογος στον τομέα των δικτύων στην κυβερνοασφάλεια με προδιαγραφές για την ασφάλεια από πλευράς της Task Force όσον αφορά πρωτόκολλα ασφάλειας για την IPSEC, πρωτόκολλα IP, επίσης στο επίπεδο του διαδικτύου ε, και των ιστοσελίδων και των ιστοτόπων μέσα στο πλαίσιο του One Web Consortium και στην κονίστρα των ε, ε, ηλεκτρονικών έχουμε τρίτης γενεάς εταιρική σχέση με την, μέσα στην οποία δραστηριοποιούμεθα με τους ομολόγους και εταίρους μας. Έχουμε επίσης και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Πώς δηλαδή οικοδομείται και χρησιμοποιείται ένα τέτοιο δίκτυο μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ποιες διεργασίες και διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των στοιχείων αυτών και των διεργασιών. Την διασφάλιση με ρήτρε ασφάλειας όλων αυτών των στοιχείων. Από την άλλη πλευρά έχουμε θέματα ασφάλειας υπό το πρίσμα της ε, εξέλιξης και της ε, προστασίας τους. Πώς θα γίνεται το logging, η καταχώρηση, πώς θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχων ταυτοτήτων και στοιχείων και άλλα στοιχεία ασφάλειας που θα διασφαλίζει ότι ο εντοπισμός ε, και η ταυτοποίηση θα γίνεται με τον πιο ασφαλή τρόπο. Διότι έχουμε εδώ μεγαλύτερη πηγή τέτοιων ε, προβλημάτων από ό,τι υποθέτει κανείς. Έχουμε μια ευρύτερη, ένα μεγάλο εύρος επαφών με εξαιρετική δουλειά για την ε, ασφαλή διεκπαιρέωση τέτοιων δεδομένων μέσω των επιχειρήσεων που θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να καλύπτονται από πλευράς ασφάλειας. Είναι κατανοητό ότι μπορεί κανείς να αναφερθεί στο, ε, στα κοινά κριτήρια όπως τα αποκαλούμε, με άλλα λόγια, όπου μέθοδοι για την βελτίωση της ασφάλειας ακολουθούνται για τα διάφορα στοιχεία κλειδιά αυτής της τεχνολογίας για τα συστήματα ανταλλαγής και λειτουργίας δεδομένων. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα ανθέξουν κάποια σενάρια απειλών και πώς μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει κανείς τις συσκευές του ε, διασφαλίζει αυτή την ε, πτυχή της κυβερνοασφάλειας. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτή την πτυχή της ασφάλειας. PCI, ε, διαδικασίες για το πώς μπορεί κανείς ε, να έχει διάδραση τέτοια αμφίδρομα ώστε να προστατεύονται όσοι εμπλέκονται στον τομέα των ενεργειακών, Για παράδειγμα έχουμε οργανώσεις όπως ΣΑΝ και ΣΑΝ ΕΛΕΚ που παράγουν προδιαγραφές και τυποποιημένα στοιχεία από πλευρά τους και έχουμε και την εξέταση ευρύτερων τέτοιων λοιπόν στοιχείων υπό την ευρύτερη λειτουργικότητά τους. Η θέση της έτσι και οι απόψεις ε, της έτσι όσον αφορά την οδηγία INS ποια είναι. Υποστηρίζουμε το γεγονός ότι θεωρείται στρατηγική σημασία ε, το πεδίο δράσης αυτό. Υποστηρίζουμε επίσης ε, την ε, προώθηση των θεμελιωδών πρακτικών και στοιχείων. Αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία έχουν τεράστια σημασία για την υλοποίηση των στόχων στον δικτυακό αυτό τομέα και την ασφάλεια πρέπει να αντλούμε από το ευρύτερο αυτό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Όσο ευρύτερη διάδοση έχουν αυτά τα στοιχεία, τόσο περισσότερο θα είναι διαδεδομένη η καλύτερη χρήση και περισσότερο ασφαλής χρήση αυτών των δεδομένων μία από τις πιο αξιοθαύμασες πτυχές είναι ο παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας, ανοιχτός και ελεύθερος παγκόσμιος χαρακτήρας, πράγμα που οδηγεί σε αμέγιστη χρήση και όσον αφορά και την οικονομία και τις ε, ε, κοινωνικές συνιστώσεις. Επίσης, η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια και οι προδιαγραφές πρέπει να αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα πολυσχηδή κριτήρια, καθιστώντας ε, διεθνείς τις προδιαγραφές στο μέτρο του εφικτού. Συνιστούμε την ε, εκπόνηση ασφαλούς μεθοδολογίας όσον αφορά την εκπόνηση μέσων και εργαλείων για την αξιολόγηση της έκθεσής μας σε τέτοιου είδους ε, απειλές. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα προϊόν το οποίο θα είναι ανθεκτικό σε τέτοιες απειλές και πώς θα μπορούμε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τέτοιες απειλές ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Πολλά μπορούν να γίνουν λοιπόν από τη διήθηση στοιχείων σε αυτόν τον τομέα τονίζοντας τη σπουδαιότητα να έχουμε μία μέθοδο πιστοποίησης ε, και αδειοδότησης αυτών των προϊόντων, ώστε η ασφάλεια να διασφαλίζεται στο ανώτατο επίπεδο εκάστοτε. Επίσης υπάρχει και μία λευκή βίβλος, ένα λευκό βιβλίο για την ασφάλεια, που είναι αρκετά εκτενές. Όμως ε, είναι πολύ, καλά, πολύ καλό στοιχείο εισαγωγικά ε, που ταυτοποιεί και προσφέρει εξοικείωση και με έναν πίνακα κατάλογο δημοσιεύσεων και σε σχέση με την βιβλιογραφία, ολόκληρη βιβλιοθήκη που υπάρχει όσον αφορά τις προδιαγραφές για την κυβερνοασφάλεια και με όλα τα στοιχεία αναφοράς που εμπεριέχονται σε αυτή τη βάση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. It's always a pleasure. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε τακτικός επισκέπτης. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή μας. Ε, σας τον παρουσίασα προηγουμένως εντάχει. Φλόριαν Walter είναι ένας ε, ανεξάρτητος σύμβουλος για θέματα ε, πληροφορικής. Είναι penetration tester έτσι ε, παρουσιάζεται ο ίδιος. Θα μπορέσει λοιπόν να μας δώσει πολλά στοιχεία. Σε 10 λεπτά ελπίζω να μπορείτε ε, να μας, πείτε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Όπως γνωρίζετε, λέγομαι Florian Walter, είμαι Γερμανός, είμαι μέλος του Chaos Computing Club. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ ως εμπειρογνώμονας, ε, απλώς σας ενημερώνω. Κοιτάξτε, το να θέλει κανείς να κάνει κάτι δεν σημαίνει ότι το κάνει και αυτό είναι το πρόβλημα της ασφάλειας του διαδικτύου από πρακτική απόξεω. Ε, ας ε, μπω κατευθείαν στο ψητό. Δεν μου δίνει σημασία η τεχνολογία. Δεν με υπακούει η τεχνολογία. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, ε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι τις μεγάλες επιθέσεις, δηλαδή στα κεντρικά, στο κεντρικό νευρικό σύστημα ε, του διαδικτύου. Είναι σαν ε, να ε, επιτίθεται κανείς στο DNA ενός ανθρώπου. Είχαμε τέτοιου είδους στο παρελθόν προβλήματα. Εκμετάλλευση των συστημάτων, για παράδειγμα συστημάτων τύπου Android, ε, όπως επίσης ε, και DDoS ε, επιθέσεις σαν αυτές που έπληξαν την Εστονία. Αυτά είναι τα σενάρια ε, για τα οποία μιλούμε, αυτά είναι τα σενάρια επί των οποίων χρειαζόμαστε συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, δεν ε, μιλάμε ότι κάποιος θα κάνει ένα, ένα ότι κάποιος θα χακάρει τον υπολογιστή ενός άλλου. για παράδειγμα, Για παράδειγμα, οι απειλές τύπου Configure. Ο ιός ε, που ήταν υπεύθυνο για αυτό το πρόβλημα ήταν ε, τόσο σημαντικός ότι ολόκληρο την υποδομή του ίντερνετ ουσιαστικά ε, την έπληξε. Ε, κόντεψε να αφανίσει το ίντερνετ. Ε, υπήρχε μια ομάδα εργασίας ε, που ονομάστηκε Conficker από τους ειδικού δικτύου του malware όπως επίσης και με ειδικού του FBI. Άλλοι εμπειρογνώμονες προσπάθησαν να συνεργαστούν για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτήν την απειλή. Αυτό που μπορούμε να δούμε λοιπόν σε αυτό αυτό το παράδειγμα είναι ότι χρειάζεται να υπάρχουν ομάδες υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, από την κοινωνία των πολιτών, από τις κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ενδεχομένως από κάθε είδους οργανώσεις που πρέπει όλοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να έχουν τουλάχιστον μία δυνατότητα να καταπολεμήσουν ε, μία τόσο τεράστια απειλή για το διαδίκτυο. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ε, μπορούμε να πάμε με πάρα πολύ συγκεκριμένο ε, σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθεί κανείς. Νομίζω ότι σε, ένα, μια πραγματικά επίγουσα κατάσταση όπως την περίπτωση Κονφίκερ δεν θα βοηθήσουν και πάρα πολύ αυτού του είδους τα μέτρα. Περισσότερο θα είναι ε, βάρος για όλους όσους θέλουν να μας βοηθήσουν να ε, μετριάσουμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, τι προτείνει ε, το ε, κείμενο που έχουμε να εξετάσουμε όλους, ε, όλες οι χώρες πρέπει να έχουν ε, επαρκώς ε, κατηρτισμένο προσωπικό για να μπορεί να αντιμετωπίσει ε, τέτοιου είδους προβλήματα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται για να διαχειρίζονται τα περιστατικά. ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συμμετέχει επίσης, γιατί τα περισσότερα συστήματα είναι ιδιωτικά συστήματα που τα διαχειρίζονται όχι κυβερνήσεις αλλά ιδιωτικοί φορείς. Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συνεργάζονται μαζί μας διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία ε, του σχεδίου της πρότασης. Συνεργασία, εκπαίδευση, κατηρτισμένο προσωπικό, με κατάλληλες δεξιότητες. Ε, όλα αυτά είναι πολύ καλά πράγματα, όπως επίσης και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν επαρκή προπολογισμό για την ανάπτυξη ένα καλό, ενός καλού ε, ΣΕΡΤ. Ενό καλού τέτοιου ε, προγράμματος αντιμετώπισης. Σε πολλές χώρες ε, συνεργάζονται με άλλες χώρες ε, πολύ καλά, Άλλες χώρες όμως δεν συνεργάζονται και ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν αυτές τις ικανότητες ε, κάποια κράτη-μέλη ε, είναι επίσης οικονομικός εν μέρη. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα χρήματα και για τα φτωχότερα κράτη-μέλη που δεν είναι δυνατόν να έχουν τέτοιου είδους υποδομές ε, και το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρογνωμοσύνης που έχει η Σουηδία και η Γερμανία για παράδειγμα. Πρέπει να έχουμε πυρογνώμονε ε, από τους ακαδημαϊκού κύκλους, ε, από όλους τους τομεί, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στα πιο περίπλοκα στοιχεία της πρότασης κατά τη γνώμη μου. Εμπιστευτικό δίκτυο κρατών μελών, ε, φορέων, οργανισμών και εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν είμαι βέβαιος ε, ότι αυτό το απόρριτο, αυτή η εμπιστευτικότητα θα βοηθήσει στη ε, συνεργασία, στην εμπιστοσύνη και όπως ακούσετε η εμπιστοσύνη είναι ένας βασικός παράγοντας εμπιστοσύνης εν προκειμένου. Το να μεταφέρει κανείς προσωπικά δεδομένα σε άλλες οργανώσεις και χώρες. Και αυτό ε, έχω κάποιους ενδιασμούς τέλος πάντων ως προς αυτό. Αλλά τέλος πάντων το πιο αστείο τέλος πάντων το χειρότερο, είναι αυτές ε, οι πληροφορίες ε, για το πόσο τροτός είναι κάποιος ε, να θεωρούνται εμπιστευτικές, να, να, να θεωρούνται εμπιστευτικές δεν νομίζω ότι το απόρριτο θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Αν δεν γνωρίζει κανείς κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Ε, πρέπει να μπορεί κανείς να βοηθήσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο όσους συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό το απόρριτο. Ε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ε, που ενδεχομένως δεν θέλει κάποιος να δημοσιεύσει ή ότι αν, δημοσιευτούν αυτές οι πληροφορίες μπορεί να βοηθήσουν ε, ε, τον ε, επιτιθέμενο. Οπότε, εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχθώ, αλλά πάση περιπτώσει αυτή η ιδέα του να υπάρξει ένα εμπόδιο εμπιστευτικότητα δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αντιθέτω, νομίζω ότι θα περιορίσει την εμπιστοσύνη τη κοινωνία των πολιτών και θα περιορίσει και την αποτελεσματικότητα του συστήματό μα. Το χειρότερο, το χειρότερο κατά την άποψή μου, είναι αυτό εδώ, ότι για να διατηρηθούν ε, οι πληροφορίες απολύτως εμπιστευτικές ε, πριν από την ε, δημοσίευση επιδιορθώσεων, τι θα γίνει όμως αν δεν επιδιορθωθεί κάτι, αν δεν, υπάρχει, αν, δεν υπάρξει διόρθωση του προβλήματος, τι θα κάνουμε. Αυτό συμβαίνει, δεν σας το λέω από το κεφάλι μου οι εταιρείες πτωχεύουν, ε, ε, υπάρχουν χιλιάδες σερβερς, αλλά μπορεί να μην υπάρχει πια η εταιρεία. Ε, έχουμε τεράστιους λόγους να πιστεύουμε ότι συχνά ε, τα προβλήματα σχεδιασμού δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα σε μία-δύο εβδομάδε. Μερικέ φορέ ούτε σε ένα μήνα δεν μπορούν να διορθωθούν. Οπότε, τι θα γίνει αν ε, αυτό που, ε, που, προμηθεύει αυτέ τι υπηρεσίε είναι ε, κάποιο ο οποίο ε, ε, σου πει κάνω ό,τι καταλαβαίνει. Εγώ δεν πρόκειται να σε βοηθήσω. Θα κρατήσω τι δικέ μου, μου πληροφορίες πάντοτε πιστευτικές Έχουμε τα στοιχεία μας ε, για την τροτότητα του συστήματός μας, αλλά δεν πρόκειται να σας το γνωσοποιήσω γιατί τα κρατάω εμπιστευτικά. Όχι. Εγώ λέω το αντίθετο. Πρέπει να δημοσιεύονται αν δεν υπάρχει κάποιος προμηθευτής ή αν ο προμηθευτής δεν θέλει να επιδιορθώσει, αν δεν υπάρχει ε, σε άμεσο χρονικό διάστημα επιδιόρθωση. Ε, μπορεί να μπορούμε να βρούμε κάποιες παρεκκλήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε πάντα κάτι να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο επικίνδυνο από το νομίζει κανείς ότι είναι ασφαλής και να μην είναι. Ε, σαν να πηγαίνει κανείς με ένα αυτοκίνητο, ε, δεν έχει φρένα και δεν το ξέρει, ενώ ε, μπορεί να είναι κανείς σε ένα αυτοκίνητο που δεν δουλεύουν ε, τα φρένα και να το ξέρει, οπότε παίρνει τις προφυλάξεις του να οδηγεί πιο αργά, για να το πω με αυτό το παράδειγμα. Ε, να δώσουμε στον προμηθευτή λοιπόν ε, μια δυνατότητα να το επιδιορθώσει. Αν όμως δεν πρέπει όμως να κρατάμε πιστευτικέ πληροφορίε, αν αυτός δεν το κάνει ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι για να ε, διατηρείται μυστικό, να διατηρείται κάτι μυστικό για πάντα. Χρειάζονται λοιπόν οι προμηθευτές ε, κάποιο ε, χρόνο, λέτε, ε, ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσετε ευθύς εξ αρχής στην πρόταση. Υπάρχουν επίσης κάποια άλλα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη μου απουσιάζουν. Πρώτον, μία ε, επαφή ε, ασφαλείας ε, δημόσια. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Αν έχει κανείς ένα RFC 2142 που είναι, χρολογείται πάνω από δεκαετία ας πούμε, αναφέρεται ότι κάθε ιστότοπος και κάθε domain πρέπει να λέει ότι πρέπει κανείς να έρθει σε επαφή με το Security at και το όνομα του domain, γιατί διαφορετικά ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ενδεχομένως αυτό το, αυτή η πρόταση να είναι ένα καλό σημείο να το εισαγάγει κανείς αυτό και να το καθαστήσει υποχρέωση για όλους να υπάρχει μια τέτοιου είδους διεύθυνση ε, στον ιστότοπο. Έχουμε επίσης το άρθρο 14.4 ε, που λέει Συγγνώμη, μπορείτε να το ξαναπάτε πίσω στη διαφάνεια. Article 14, 4. Το άρθρο 14.4 λοιπόν, όπου λέει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να ενημερώνει το κοινό αν το περιστατικό είναι δημόσιου ενδιαφέροντος. Μπορεί, πρέπει δεν είναι κάτι το δυνητικό, είναι κάτι το υποχρεωτικό. Πρέπει να ενημερώνεται ε, το κοινό. Προς τα μπροστά θέλω να πηγαίνουν οι διαφάνειες και όχι προς τα πίσω. Άρθρο 13. Ε, Τέτοιε συμφωνίε θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς προστασίας προσωπικών δεδομένων που ε, ε, υπάρχουν στο δίκτυο συνεργασίας. Ε, ε, ναι, ίσως, όχι. Το άρθρο 15, σημεία 2 και 3, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιες εταιρείες να περάσουν έλεγχο ασφαλείας. Εντάξει, δεν λέω, αλλά για ποιο λόγο και κάποιες θα έπρεπε να υποχρεώνονται να περνούν έναν έλεγχο ασφαλείας και θα έπρεπε να παίρνουν και τις απαραίτητες ε, προφυλάξεις ε, και τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Ε, κάτι τέτοιο μπορεί να στοιχήσει πάρα πολύ ένας τέτοιος έλεγχος. Ποιο θα το πληρώσει αυτό. Αν αυτό επιβάλλεται σε μία μικρή εταιρεία τρει φορές το χρόνο, θα πτωχεύσει η εταιρεία. Οπότε εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά βάλτε κάποια όρια τουλάχιστον για μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές ε, οι οδηγίες, ε, οι υποχρεώσεις ε, πρέπει να μπορούν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο. Δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσουμε τον κόσμο να κάνει έλεγχο ασφαλείας να... και να μην μπορεί κανείς να κάνει τίποτε αν κάτι δεν πήγε καλά. Επόμενη διαφάνεια. Αυτό το είπα ήδη, επόμενη διαφάνεια. Ε, επίσης κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν αναφέρεται, το είπε προηγουμένως ε, η Εστονή συνάδελφος, ε, η παροχή ύδατος, το, η πιο κρίσιμη υποδομή για όλους. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο πρότασης. Εσείς πιστεύετε ότι τώρα το νερό έρχεται στις βρύσεις μας χωρίς υπολογιστές. Αν λάθος κάνετε, γιατί λοιπόν τα τρόφιμα και το νερό δεν καλύπτονται. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πρώτο σε περίπτωση καταστροφής. Χρειαζόμαστε Χρειαζόμαστε το νερό. Χρειαζόμαστε τα τρόφιμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much uh, for... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ξεκάθαρη παρουσίασή σας. Έχετε εμπλακεί σε πολλούς τομείς. Αυτό που έχω σήμερα για τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. Will Sample θα μας δώσει την άποψη κάποιου που έχει εμπλακεί εις βάθος σε έναν μεγάλο οργανισμό που εξαρτάται απόλυτα από τους υπολογιστές και την πληροφορική. Η Σάντρα θα σας βοηθήσει με την τεχνολογία. Δουλεύει τώρα, έτσι. Good afternoon. Thank you, Chair. Καλησπέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Will Sample με λένε και αντιπροσωπεύω το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ομάδα μου είναι η ομάδα διαχείρισης απειλών και ευαλωτότητας πριν από τέσσερα χρόνια δημιουργήθηκε μετά την εξέλιξη των κυβερνοεπιθέσεων και των κοινοπηλών που αντιμετώπιζε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ αλλά στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλη παρουσία και στην Ευρώπη και στην Ασία. Είμαστε Έχω δεχόμαστε τι περισσότερες επιθέσεις. Ο χρηματιστικό θεσμό που δέχεται τι περισσότερες υποθέσεις στον κόσμο. Και η γραμμή μου είναι στην πρώτη γραμμή, προσπαθεί να μειώνει και να αποφεύγει και να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις. Και εγώ θα μιλήσω για την ε, οδηγία για την προστασία των δικτύων και να αναφερθώ τι κάνουμε ήδη εμείς σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, διάχυση πληροφοριών είναι απειλές όσον αφορά την ομάδα μας διαχείριση της ευαλωτότητας είναι θέμα διατύπωσης γλώσσας, συνεργασίας, ορισμού. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε από παλιά είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή γλώσσα για να μπορούμε να επικοινωνούμε με εταίρους μας και σε όλους τους ε, θεσμούς σχηματοπιστωτικούς και να επικοινωνούμε και με τις υπηρεσίε ασφαλείας και αστυνομία των χωρών στις οποίες δρούμε, δραστηριοποιηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό, μάθαμε επίσης, ότι δεν υπήρχαν κοινά πρότυπα ε, γινόταν πολλή δουλειά αλλά τίποτα δεν είχε επισημοποιηθεί και όλοι θεώρησαν ότι οι κυβερναπηλές ήταν κάτι διαφορετικό. Ένα από τα πρώτα πράγματα που προσπαθήσαμε να κάνουμε εντός της ομάδας εργασίας μας, σηματοστατικές υπηρεσίες, να καθορίσουμε τις κυβερναπηλές και να καθορίσουμε πώς και τι μοιραζόμαστε. Αυτοί οι ορισμοί που αναφέρονται στο άθρο 3 είναι σημαντικότατοι. Πρόκληση που αντιμετωπίσαμε πώς να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τις ε, πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών εις απειλές στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται περί πληροφορίες μυστικές, τέτοιου είδους. Αν μοιραζόμαστε ε, μεταξύ οργανισμών και χωρών ε, πληροφορίες για απειλές, είναι απόρριτες πληροφορίες. Μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε απειλή, η πρόθεση να απειλήσουν ένα οργανισμό ή μπορούμε να κοινοποιήσουμε την απειλή προς έναν οργανισμό ή μια χώρα. Τώρα η κατανάλωση των πληροφοριών, τυποποίηση των πληροφοριών αυτό και η κοινοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τι απειλέ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ξεκινάμε να προχωράμε όσον αφορά την αντιμετώπιση τη διαχείριση των κυβερναπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ε, μπορούμε να ερμηνεύουμε σωστά, με κεραιότητα και με πιστότητε πληροφορίε. Τι μάθαμε εμεί στο ταξίδι μα, ότι δεν είναι όλε οι πληροφορίε καλέ. Πρέπει να ξεψαχνίζουμε τι πληροφορίε. Να δούμε ότι οι πληροφορίε που λάβαμε πραγματικά έχουν επαληθευτεί, έχουν εξεταστεί. Διαφορετικά τελικά ξοδεύουμε χρόνο, πόρους, κύκλους επιβεβαιώνοντας κατά πόσο οι πληροφορίες αληθεύουν είτε όχι. Και ένα ιδιωτικό φορέα αυτό σημαίνει δαπάνες. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε την πρόθεση εκείνων που διαπράττουν την απειλή, εκείνων που απειλούν. Αυτοί προσπαθούν να επιτεθούν στις υποδομές μας. Δεν άκουσα να αναφέρεται μέχρι τώρα ή σε σχέση με την οδηγία τίποτα όσον αφορά την κατανόηση των κινήτρων, της συμπεριφοράς, πρόθεση των επιτιθεμένων. Γιατί επιτίθεται αυτός ο κόσμος κατά των κρισίμων μας υποδομών. Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Κάνουμε ανταλλαγέ πληροφοριών, πραγματοποιούμε ανταλλαγέ πληροφοριών, υιοθετήσαμε κάποιε από τι πρακτικέ που χρησιμοποιούνται. Sticks, ε, βλέπετε, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που λάβαμε για να ετοιμάσουμε, να πληροφορήσουμε το κέντρο επιχειρήσεων. Καταναλώνουμε δηλαδή τα στοιχεία που δεχόμαστε και παράγουμε, προσαρμόζουμε τα μέτρα μείωσης και αντιμετώπιση του κινδύνου δεόντος. Επίσης θέλουμε να καταλάβουμε πολύ καλά ποια είναι τα κίνητρα εκείνο που διαπράττουν αυτές τις πράξεις. Θα ακούσατε τις ειδήσει να αναφερόμαστε με τους ανώνυμους. Ε, εμάς κυνηγάνε πρώτα οι ανώνυμους διότι είμαστε κεφαλοκική πρωτεύουσα του κόσμου και είμαστε μεγάλος στόχος. Ε, ε, θέλουμε να καταλάβουμε γιατί αυτοί κινούνται έτσι και πώς μπορούμε να μειώσουμε τα αποτελέσματα των επιθέσεων και τις απειλές που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε θέλουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις απειλές. Το δίκτυο διάχυσης πληροφοριών, διάχυσης πληροφοριών θα πρέπει να ασχολείται με την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα οργανισμών και στα επίπεδα, στα επίπεδα διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων πολυεθνικών. Και πρέπει να μπορούμε να προσμετρήσουμε τον κίνδυνο, την απειλή και αυτή είναι πολύ δύσκολη έννοια. Διότι η απειλή για το κάθε οργανισμό σημαίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό είναι σημαντικά τα πρότυπα. Αν μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον κάποια μορφή προτύπων, προδιαγραφών που να μπορούμε να μετρήσουμε την απειλή, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα μείωση των αποτελεσμάτων του κινδύνου και αντιμετώπιση των κινδύνων και να βοηθήσουμε και άλλου οργανισμού που δεν είναι τόσο ικανοί να αντιμετώπισουν τον κίνδυνο και είναι καθοδόν προ την ανάπτυξη μέτρων αντιμετώπιση. Θέλουμε να κινηθούμε από κίνδυνο σε απειλή. Δεν επιτιθέμεθα κατά εκείνων που ακολουθούν την προσέγγιση του κινδύνου, αλλάζουμε το είδο τη προσέγγιση. Ο κίνδυνο καλό είναι προ προσέγγιση, αλλά υπάρχει απειλή, είναι παρούσα και όλε οι αντιμετωπίσει μέσα στον κίνδυνο δεν ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή. Οι αξιολογήσει των κινδύνων είναι το μυστικό όπλο του επιτιθεμένου. Και αυτό είναι πρόβλημα του ιδιωτικού τομέα κυρίω. Μπορούμε να διενεργούμε αξιολογήσει κινδύνων στην οργάνωσή μα, μπορούμε να δεχτούμε τον κίνδυνο επίση. Αυτό είναι πρόβλημα. Η απειλή δεν ασχολείται με, τον, με την αποδοχή του κινδύνου, εκμεταλλεύεται τον κίνδυνο η απειλή. Είναι επιχειρησιακή κίνδυνη και όχι στρατηγική, είναι τακτική φύσεω. Επιχειρησιακή καθημερινά βρίσκονται απειλέ. Ε, δεν θα φύγουν ανάλογα με το πότε είναι η επιχείρηση ενωμένη με το διαδίκτυο. Ε, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί απειλή, όχι τόσο. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται ε, διάδοση πληροφοριών. Άρα πρόκειται περί επιλογής. Με τους κίνδυνους έχει την επιλογή. Δέχεσαι τον κίνδυνο, δεν το δέχεσαι. Με την απειλή σου έρχεται η απειλή ανεξάρτητα με αυτό που θες εσύ. Θες δεν τη θες, σου έρχεται η απειλή. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από κάποιον που θέλει να μας απειλήσει. Δεν μπορεί να κρυφτείτε από, το... μπορεί να κρυφτείτε από τον κίνδυνο. Ε, συμπεριέλαβα κάποιους ορισμούς κινδύνου και απειλών. Με την ησυχία σας μετά μπορείτε να τα δείτε. Οι διαφάνειες μπορούν να κατέβουν το διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορίε. Χρειάζεται μια σωστή αντιμετώπιση του κινδύνου. Και ο ιδιωτικό και ο δημοσιοτομέα θα μπορούν να ετοιμάσουν σχέδια προβλέψιμα για να αντιμετωπίσουν τις προθέσεις ομάδων που θέλουν να επιτεθούν κατά κρισίμων εθνικών υποδομών και να βλάψουν την οικονομία. Αν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες, βελτιωνόμαστε, δυναμώνουμε. Έχουμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε μικρές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να προξενήσουν πολύ μεγάλες ζημιές σε εταιρείε και εταιρικέ υποδομές και εθνικές υποδομές. Θέλω να μειώσουμε τις δυνατότητες που έχουν με το μοίρασμα των πληροφοριών σε μια κοινότητα μειώνουμε τη δυνατότητα του κακού να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό σημαίνει ότι αν μοιραστούμε και συνεργαστούμε όσον αφορά τις πληροφορίες που διαθέτουμε, μειώνουμε τη δυνατότητα των επιτιθέμενων να πετύχουν το σκοπό τους. Πρόληψη είναι ευκαιρία. Άρα η απειλή απ' έξω γίνεται ευκαιρία για την κοινότητα. Ισχυροποιούμε με την Ένωση. Λοιπόν, απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής. Απά, ε, διαφάνεια, ε, μπορεί να βλαφτεί μια εταιρεία, πνευματικά δικαιώματα, όλα τα επιχειρήματα του ιδιωτικού τομέα. Είναι επιχειρήματα του ιδιωτικού τομέα να μην διαδίδει πληροφορίε. Είδαμε στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη ότι ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Αν μοιραζόμαστε πληροφορίες εντός του χρηματοστατικού τομέα, βοηθάμε ε, την κοινότητα. Δεν δίνουμε ανταγωνιστικό όφελος, ε, ισχυροποιείται η αγορά. Πρέπει να δούμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής με σχετικά μέτρα. Θέλουμε να έχουμε κάποια σημάδια, σημεία που δημιουργούν εμπιστοσύνη. Και δεν θέλουμε να προσφεύγουμε πολύ συχνά σε αυτό. Εμείς ρυθμιζόμαστε πολύ αυστηρά σαν ε, χρηματοστατικό ίδρυμα τέτοιου μεγέθους. Δεν χρειαζόμαστε ε, δικαιολογίες για να φαινόμαστε καλοί και να μπει το κακό, η κακή φήμα δημιουργηθεί από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, ε, επιλεκτική, επιλεκτικό μοίρασμα, υιοθέτηση μέτρων καθυστερισμένα, μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι αρνητικά στοιχεία που μπορούν να συμβούν εάν δεν εξετάσουμε τις δυνατότητες ε, να δίνονται πληροφορίες θέλουμε να δημιουργήσουμε ελέγχου που επιτρέπουν προστασία ιδιωτική ζωή. Θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί για την κοινότητα και όχι βάρο. Χρειάζεται συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένη μορφή και να ξέρει αυτός που είναι τις πληροφορίες τι μπορεί να σημαίνει κακή χρήση των πληροφοριών. Αυτή θα είναι η επιτυχία, αν καταλάβουν οι εταιρείε τελικά τι διακυβεύεται, αν δίνουν ή δεν δίνουν πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Ήταν πολύ επικοδομητικό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για τους ε, συντονιστές, για τις συνεδρίες των συντονιστών. Εφόσον εδώ δύο συντονιστές, δεν θα τους νοιάζει να παρατείνουμε λίγο αυτή τη συνεδρίαση. Ο κύριος Σβάμπ θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Και στο Ζιζέπε Αλμόντε θα ήθελα να δώσω και την ευκαιρία να πει κάτι. Σίγουρα κράτησε πολλές σημειώσεις και θα θέσει ερωτήσεις στους ομιλητές. Άντρια Σβάμπ, έχεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θες να θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά μετά από αυτές τις τέσσερις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων υπάρχουν πολλές αντιφάσεις, πολλά ερωτήματα και ερωτηματικά που δεν, δεν μπορώ να τα διατυπώσω όλα. Σε δύο θα επικεντρωθώ. Το ένα η παρατήρηση του κυρίου Σάμιουσεν που σε σχέση με τον ορισμό των κέριων υποδομών τοποθετούμενος είπε η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λέει υπερβολικά ευρεία αυτό κάπως αντιφάσκει σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βάλτερ, ο οποίος ρητά αναφέρθηκε στην υδροδότηση στη Γερμανία, στην γερμανική υδροδότηση είπατε δεν θέλετε να εμπλακείτε. Αυτό όμως ως σχόλιο εν παρόδο το επιχείρημά σα όμω μετά από μια πρώτη ματιά μπορώ να το δεχτώ. Το θέμα είναι στο τέλο τέλο ποια είναι η κέρια και κύρια υποδομή. Υπάρχουν κάποιε αντιφάσει ακόμα αλλά όχι κάποια κύρια λύση. Ίσως κάποιο πραγματογνωμονο μπορεί να με βοηθήσει να βρούμε αυτή τη λύση. Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω ή παρατηρήσω είναι το εξή. Καταρχήν θέλουμε με την οδηγία αυτή την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αγορά να την αυξήσουμε. Θέλουμε ένα μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας για πιθανές διαρροές, για πιθανές επιθέσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το ασφαλέστερο πλαίσιο, αλλά με έναν τρόπο που θα ενθαρρύνει στη συνεργασία και δεν θα αποτρέπει ή αποθαρρύνει στη συνεργασία. Και είπατε ότι με κανένα τρόπο λέει δεν θέλετε να παρακρατούνται πληροφορίες. Προκλητικά το αναφέρετε αυτό στη διατύπωσή σας έτσι ή πράγματι εννοείται ότι οι πληροφορίες για διαρροές είναι κέρδος για όλους που οπωσδήποτε θα έπρεπε να διαχέονται αυτές σε σχέση με τις γενικές πληροφορίες που θα ε, επιλέγατε έναντι οποιασδήποτε σκέψης ε, του τι θα έπρεπε οποτεδήποτε ήδη να είναι διαθέσιμο για την εξέβρεση λύσεων. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις, Πρόεδρε, δεν θα υπάρχει χρόνος για περισσότερα. Ε, um, Καλώς. Άλλος συνάδελφος. Έχει άλλες ερωτήσεις. Τζουζέπε, θες να μιλήσεις. Έχεις ερωτήσεις. Ή θες να συνοψίσεις το τέλος. Ο Γκιουζέπε να μας πει κάτι. Και μετά να δώσω ένα λεπτό στον καθένα από τους εμπειρογνώμονες να συνοψίσει. Ο Γκιουζέπε, πρόεδρε, τέσσερα πράγματα να πω αν επιτρέπετε. την άδειά σα, τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Πολλά περισσότερα θα ήθελα να πω, αλλά σε τέσσερα θα επικεντρωθώ. Στο πρώτο θέμα, είπατε ρωτήθηκε το προκλητικό ερώτημα. Μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα της εμπιστοσύνης. Όχι, αλλά μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία για την προώθηση αυτής της ε, ε, εμπιστοσύνης και στην ε, δειγματοληπτικά από πλευράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας υπάρχει συνεργασία για την προώθηση εμπιστοσύνης από τους εμπλεκόμενους, για τη διασφάλιση αυτής της συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσω, στη, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα παραδείγματα, η ρύθμιση, η συνεργασία όσον αφορά τις απαιτήσει για τις ε, δημόσιες ε, υπηρεσίες, ε, για παράδειγμα για την διασφάλιση της τροφοδότησης με φυσικό αέριο, η συνεργασία στο πεδίο της υγείας, ώστε διασυνοριακά να μπορούμε να επαρκέσουμε. Ξέρουμε ότι η εσωτερική αγορά σε σχέση με, το, με την νομική βάση υπάρχουν απαιτήσει που υφίστανται για τη συνεργασία αυτή διασυνοριακά και σε κάποιους τομείς ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζετε έχετε εξοικειωθεί με αυτό δηλαδή προστασία καταναλωτών κυρίως συνεργασία σε δίκτυα για την προστασία καταναλωτών πράγμα που απαιτεί έναν φορέα μια υπηρεσία για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων ή παραβάσεων ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται τέτοιου είδους ε, ε, διώξεις ή κυρώσεις ε, διασυνοριακά όταν υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια στοιχεία επαρκώς. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι Πολλά μπορούν να αναφερθούν για τα όρια της εθελούσιας προσέγγισης που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα. Ο κύριος περιοριστικός όμως παράγοντας είναι ο αποκλεισμό. Με άλλα λόγια το γεγονός ότι κάποιοι αποκλείονται. Το δυναμικό για παράδειγμα που δημιουργείται, το εθνικό δυναμικό είναι μια προϋπόθεση για να υπάρξει εμπιστοσύνη και να εμπλέκεται κανείς ισότιμα με άλλους σε ένα τέτοιο φορέα. Αυτή τη στιγμή δεκα κράτη-μέλη υπάρχουν που κάποια από αυτά, και αυτό δεν, είναι, δεν εκπλήσει κανένα, υπάρχουν και ανάμεικτα συναισθήματα όσον αφορά την οδηγία αυτή σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται γύρω από αυτή την τράπεζα Τώρα, σε σχέση με την πλειοψηφία, 17 ή 18 κράτη-μέλη αποκλείονται από αυτή τη συνεργασία. Και αυτό όσον αφορά την λειτουργία αυτή που αφορά μια συνολική πανευρωπαϊκή προσέγγιση και δράση, οι πιο δύναμη κρίκοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευση προζημίαν συνολικά των υπόλοιπων. Έγινε πολλής λόγος λοιπόν για το τι διακυβεύεται εδώ και τις απαιτήσει ε, για όσους εμπλέκονται στις αγορές και τις ε, δημόσιες αρχές, τις υποχρεώσεις που υφίστανται ώστε να υπάρξει ένας τέτοιος ε, ευρύτερα αποτελεσματικός πολιτισμός για την ασφάλεια. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι εχθές είχαμε την πρώτη συνάντηση για το, την πλατφόρμα ε, ασφάλειας δικτύου που θα είναι μια ΣΔΙΤ, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τις βέλτιστες πρακτικές από τις οποίες πρέπει να αντλώνται από τις διεθνείς προδιαγραφές ε, και επίσης κίνητρα που πρέπει να δίδονται ώστε να ενθαρρυνθεί και να προτρέπεται η υιοθέτηση τέτοιων προδιαγραφών όσον αφορά τους εμπλεκόμενους και τις ε, δημόσιες αρχές από πλευράς ε, κρατών. Και τέλος και κάτι άλλο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι και προτιμώ να μην αναφερθώ στο ε, εδάφιο εκείνο σε σχέση με την δημοσιοποίηση συμβάντων και στοιχείων. Αλλά αυτά τα οποία εν συντομία έχουμε ε, ακούσει από τη βιομηχανία, δηλαδή για το ευάλωτο του χαρακτήρα στο ε, λογισμικό, στο hardware ή στο software, είναι κάτι το οποίο συνολικά θα εξισωνόταν με τη δημιουργία στόχου, στοχοθέτηση των υπηρεσιών αυτών που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο software ή hardware, με άλλα λόγια. Και τέλος, δεν θα έπρεπε να υπερεκτιμούμε το κόστος όλων αυτών που κάνουμε. Θα πρέπει να είναι αναλογικό το κόστος αυτός και αυτό και όχι υπερβολικό. Θα πρέπει το δυνατόν περισσότερο να μπορέσουμε από πλευράς μελέτης επιπτώσεων να κρατήσουμε στα όρια αυτό το κόστος. Και από πλευράς εκτιμήσεων που είναι σημαντικό να υπάρχουν και εκτιμήσεις σε σχέση με την οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες, από ό,τι θα γνωρίζετε, οι αρχές αρμόδιες για τις ε, τηλεπικοινωνίες ε, πρέπει να έχουν ε, εντάξει τις, την έκθεση στους κινδύνους στις εκθέσεις τους. Βασιζόμενοι σε αυτά τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός τέτοιων συμβάντων ετήσια θα πρέπει να είναι 1.700 τέτοιες περιπτώσεις. Από αυτές τις 1.700 μόνο 150 ή 250 διασυνοριακά είναι εκείνες που αναμένονται ότι θα τύχουν ε, σε βάθος εξέτασης πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι τόσο ε, μεγάλο, τόσο ε, βαρύνο στοιχείο και πιστεύουμε ότι το κόστος το οποίο θα απορρέει για τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι πραγματικά αναλογικό και θα μπορούν να το επομισθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που απαντήσατε πιο συγκεκριμένα και σε άλλα σημεία. Θα κάνουμε το εξή. Να καλέσω τον καθένα από του ομιλητέ να δώσει μια γρήγορη απάντηση στις ερωτήσει του κ. Βάμπ και να πούνε τι άλλο θέλουν. Ο κ. Σέμπλ να ξεκινήσει. Και θα ακολουθήσουμε τα διάφορα μέλη του πάνελ και αν κάποιοι από τα μέλη του πρώτου πάνελ θέλουν να πούν κάτι μπορούν να προσεκίσουν την προσοχή. Ο κύριος Σέμπλ πρώτα απ' όλα. Πολλές αντιφάσεις υπάρχουν όσον αφορά τις πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν πολλές απόψεις και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να έχουμε αυτή την άποψη. Από τη μία πλευρά είναι πολύ καλό να λέμε ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά την υποβολή αναφορών και ευάλωτων σημείων για προϊόντα και υπηρεσίες Απ' την άλλη είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Ε, πρέπει να υπάρχει μέση και ισορροπία και εξαρτάται για κάθε συμβάν και πρέπει να πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές οι οργανισμοί θα επιτρέψουν να συνεχίζεται μια επίθεση για να μαζέψουν περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουν τα στοιχεία αυτά να υποστηρίξουν καλύτερες ανταποκρίσεις για άλλους, άλλους φορείς και για να βοηθήσουν αυτά τα στοιχεία για ειδήποτε νομική δίωξη μπορεί να ακολουθήσει. Είναι σωστές αυτές οι απόψεις, αλλά ανάλογα ποικίλουν οι απόψεις αυτές ανάλογα με το συμβάν. Ευχαριστώ, ναι. Αυτή η δημοσίευση στοιχείων για ευάλωτα σημεία δεν ήταν κάτι αστείο. Σοβαρά το εννοούσα όχι κάθε φορά πριν να υπάρξει διορθωτικό μέτρο. Αν ανακαλύψετε ότι υπάρχει ένα κενό και, και δώσετε χρόνο στον πολιτή να το φτιάξει και θέλει να το φτιάξει ο πολιτής και είναι συνεργάσιμος και κάνει ό,τι πρέπει για να διορθωθεί η κατάσταση, μετά αφού γίνει η διόρθωση πρέπει να δημοσιευθούν οι πληροφορίες για το ευάλωτο σημείο. Αλλιώς μόνο οι κακοί έχουν τη γνώση του πώς να εκμεταλλεύονται τη συγκεκριμένη αδυναμία. Διότι το patch που στέλνει ο πολιτής ήδη είναι μια συνταγή για εκμετάλλευση. Διότι το patch αυτό, το πρόγραμμα το μικρό για να διορθώσει το κενό, συμπεριλαμβάνει όλα όσα έχουν αλλάξει στο πρόγραμμα. Άρα ξέρεις και ποιο είναι το πρόβλημα ήταν το πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα βγει η διόρθωση, το διορθωτικό προγραμματάκι και το patch, οι πληροφορίε για το πρόβλημα ήδη έχουν δημοσιευτεί. Είναι σε γλώσσα μηχανή. Αφού βγει το patch, δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην δημοσιευθούν οι λεπτομέρειε για την αδυναμία. Οι πολιτέ δεν θέλουν να γίνεται αυτό, ε, διότι δεν είναι πολύ καλό να πει κανείς δημοσία ότι έκανα λάθος εν πρώτης και δημιούργησε πονοκεφάλους για πολλούς. Βέβαια, φυσικό αυτό, όμως πρέπει να το κάνουμε αυτό για να δώσουμε και στους πολιτές κίνητρο να γίνουν καλύτεροι όσον αφορά την κατασκευή λογισμικού και ασφαλούς λογισμικού στο μέλλον. Άρα πρέπει να έχουμε ε, υπόψη οι ειδικέ περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πολιτή. Ο πολιτής δεν είναι συνεργάσιμος κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάτς Νίλσον. Ε, μερικές παρατηρήσεις και από πλευράς μου αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλές αντιβάσεις στον τομέα αυτό και νομίζω ότι οι προθέσεις είναι οι ίδιες ε, όταν, για παράδειγμα, κυβερνητικοί φορείς ε, με, για κέρυες υποδομές ε, μπορούν να συνεργαστούν ε, για την προστασία αυτών, για ανταλλαγή πληροφοριών, για ανάλυση απειλών, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο για να αυξήσουν την ασφάλεια των δικτύων, όπως επίσης να βρούμε και τα σωστά κίνητρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δουλειά ε, η πρόθεση είναι η ίδια, αλλά ενδεχομένως κάποιοι μηχανισμοί που πρέπει να γίνουν πιο κατανοητοί είναι να πτυχθούν λίγο περισσότερο. Εμείς ε, ως προμηθευτές τεχνολογίας πρέπει να πω ε, ότι μία πιο οριοθετημένη και ασφαλής κατάσταση στην Ευρώπη θα έδινε τη δυνατότητα μικρότερου κατακαιρματισμού, εξοικονόμησης χρημάτων που δημιουργεί τέτοιου είδους καταγερματισμός, αν ο καθένας δηλαδή διαχειριζόταν με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα προβλήματα στο κράτος μέλος του, ε, εφόσον ζούμε σε μια διεθνή, ε, βρισκόμαστε ενώπιον μιας διεθνούς κατάστασης. Η συνεργασία για τα θέματα ε, πολιτικής είναι επίσης πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών ε, για ε, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Όσο ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όσο πιο πολύ συνεργαστούμε, τόσο καλύτερα μπορούν να είναι τα αποτελέσματά μας. Κύριε Σάμιουλσον, ευχαριστώ πολύ να απαντήσω κι εγώ σύντομα σε αυτά που είπε ο κύριος Φαμπ και σε αυτά που ρώτησε για τις κρίσιμες υποδομές. Νομίζω ότι η Σουηδία θα ήθελε κάποιες απαιτήσει ε, για τον ηλεκτρισμό, το αέριο και γιατί όχι και για το νερό. Ε, για τα κοινωνικά ε, δίκτυα επίσης, όλα αυτά τα όλα αυτά τα στοιχεία με τα οποία κανείς, χωρίς τα οποία κανείς δεν μπορεί να ε, ζήσει αν υπάρξει κάποια επίθεση. Επίσης, ε, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέγεθος της εταιρεία ε, από πλευράς ε, αριθμού υπαλλήλων. Μπορεί όμως να είναι λιγότεροι οι άνθρωποι που χειρίζονται ένα τεράστιο σερβερ και μπορεί να υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιος αριθμός προσωπικού για, μικρότερο, για μικρότερους σερβερ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι πραγματικά κερδίσαμε πολλά από ε, τις ομιλίες σας. Ε, ήταν άλλωστε ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Άντριου Σφάμπ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να συνοψίσουμε. Θέλεις οπωσδήποτε να πεις ε, κάτι. Αν όχι, να σε ευχαριστήσω γιατί οργάνωσες αυτήν την ε, ακρόαση. Μέχρι το τέλος ε, του Ιουνίου πρέπει να έχουμε την ε, έκθεσή σου. Αύριο το απόγευμα θα γίνει μία συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Θα πάω εγώ εκ μέρους του κυρίου Σφάμπ. μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, να δείτε στο διαδίκτυο τη συνεδρίαση αυτή. Ελπίζω μέχρι τον Νοέμβριο να έχει εγκριθεί η έκθεση, αλλά πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και Βιομηχανίας. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ξεκινήσατε τη διαδικασία. Συγγνώμη, πρέπει να σας ζητήσω να αποχωρήσετε γιατί έχουμε μία ε, συζήτηση με τους ε, συντονιστές που είναι και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν ήμασταν ιδιαίτερος φιλόξενοι, αλλά βεβαίως ευχαρίστως να συνεργαστούμε μαζί σας ε, κατά τους επόμενους μήνες.